Αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα. Ah, Δεν έχω και... Σπυράκι. Ε, ε, αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Allez, prenez place. Καθίστε παρακαλώ. Les advisors και οι σύμβουλοι Δεν έχω και το σφυράκι μου. Πολύ ωραία. Σας παρακαλώ οι σύμβουλοι του ΕΛΚ να σταματήσουν το πηγαδάκι γιατί κάνετε αρκετή φασαρία σήμερα. Θα ξεκινήσουμε παρακαλώ. Le projet d'ordre du jour. Μπορούμε να εγκρίνουμε το σχέδιο ημερήσιας διάταξη αν δεν υπάρχουν ενστάσεις. Εξακολουθείτε να κάνετε πολύ φασαρία. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ωραία, ευχαριστώ. Μπορούμε να εγκρίνουμε το σχέδιο μερισσίας διάταξης αν δεν υπάρχουν ενστάσεις. Ανακοινώσεις της Προέδρου. Στα έγγραφά σας έχετε τις αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν από τους συντονιστές ε, στη συνεδρίαση που έγινε στις 18 Ιουλίου. Οι αποφάσεις σας έχουν διανεμηθεί και είναι διαθέσιμες επίσης και στο intranet διότι είμαστε λίγο πιο οικολόγοι πλέον και χρησιμοποιούμε πληροφορική. Αυτό λέγεται e-committee. Εάν δεν υπάρχουν ενστάσεις μέχρι τις 12.30 θεωρούμε ότι εγκρίνονται οι αποφάσεις από την Επιτροπή μας. Επόμενη ανακοίνωση της Προέδρου σας που αφορά την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί την οδηγία του 2008-96 για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών. Έκθεση της κυρίας Αγιούτο. Στα έγγραφά σας θα βρείτε το κείμενο της οδηγίας για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών η Επιτροπή Μεταφορών ψήφισε στις 10 Ιανουαρίου του 2019 μετά από την εντολή της Επιτροπής Μεταφορών ε, η ομάδα διαπραγματεύσεων ε, με την εισηγήτρια τότε την κυρία Ντανιά Λαγιούτο διαπραγματεύτηκε το κείμενο με το ε, ο Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Επιτροπή μας επιβεβαίωσε την διοργανική συμφωνία που ελήφθη προσωρινά με ψηφοφορία στις 4 Μαρτίου. Εν τω μεταξύ, οι γλωσσομαθείς νομικοί οριστικοποίησαν το κείμενο και ε, υπάρχει ένα κοριγέντουμ το οποίο αντανακλά όλες τις τροποποίησεις που έγιναν μετά από την έγκριση και οι γλωσσικές αλλαγές που έγιναν στο κείμενο, οι οποίες είναι ίσονο σημασίας και απλώς ε, τεχνικές. Η καινοτομία όμως είναι ότι επειδή η κυρία Γιούτο η προηγούμενη συγγήτρια. Δεν είναι πλέον ε, ευρωβουλευτής, διότι δεν επανεξελέγει. Η διαδικασία της διόρθωσης είναι κάτι το οποίο είναι πολύ συνηθισμένο. Ε, θεωρώ λοιπόν ότι η συμφωνία εγκρίνεται, εκτός και αν υπάρχουν ενστάσεις. Ευχαριστώ και σας παρακαλώ να τις διαβιβάσετε στη γραμματεία μέχρι το τέλος της ε, ημέρας, αν υπάρχει κάποια αλλαγή για το σημείο αυτό. Έχουμε και επισκέπτες σήμερα στην αίθουσα. Να καλωσορίσω μια ομάδα φοιτητών από το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων ε, Επιστημών από τη Βεσφαλία, ε, προσκεκλημένη του κυρίου Έρτουγ. Καλωσορίσατε λοιπόν στην Επιτροπή Μεταφορών και σας παρακαλώ να παρακολουθήσετε τη συζήτηση γιατί έχουμε εδώ παρουσία της Φιλινδικής Προεδρίας. Έχουμε μία γυναίκα Υπουργό Μεταφορών και μία γυναίκα Υπουργό Τουρισμού. Μπορεί δηλαδή κάποιος να είναι γυναίκα και ταυτόχρονα να αναλαμβάνει και κομβικά υπουργεία. Ε, να τις καλωσορίσουμε και να τις χειροκροτήσουμε για την παρουσία τους εδώ. Και θα ξεκινήσουμε με την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι τιμή και χαρά για μένα να δώσω το λόγο στην κυρία Σάνα Μαρίν, η οποία είναι η Φιλανδή Υπουργό Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών, και στην κυρία Κάτρι Κουλμούνη, η οποία είναι η Φιλανδή Υπουργό Οικονομικών Υποθέσεων. Να σας καλωσορίσω λοιπόν, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στην Προεδρία σας. Όπως γνωρίζετε, η Φιλανδική Προεδρία έχει πάρα πολλές προτεραιότητες Ε, και σε αυτή την εβδομάδα είχατε και αρκετά πράγματα να κάνετε. Ε, θα έχουμε λοιπόν σήμερα την ευκαιρία να συζητήσουμε περισσότερες λεπτομέρειες ε, για τους τομείς της αρμοδιότητάς σας, να μας πείτε ποιες είναι οι προτεραιότητές σας, τι θέματα θα ε, προωθήσετε. Ε, εγώ χαίρομαι που έχουμε εδώ ε, τρεις γυναίκες που ασχολούνται με τα θέματα αυτά, διότι νομίζω ότι σήμερα υπάρχει πλέον διάθεση να δείξουμε ότι ο τομέας των μεταφορών δεν είναι ένας τομέας ο οποίος αφορά μόνο τους κυρίους, λυπάμαι για σας, αλλά ε, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και εμείς οι γυναίκες ε, στην πολιτική μεταφορών. Πρόκειται για μια τεράστια πρόκληση. Οι μεταφορές είναι το 30% των αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου. Όλοι μιλάνε για την κλιματική αλλαγή και αυτό είναι ο μόνος κλάδος ο οποίος δεν καταφέρνει να μειώσει τις εκπομπές του από το 1990. Πρέπει λοιπόν πραγματικά να φροντίσουμε ο τομέας αυτός ε, να... Ε, μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτή την τεράστια πρόκληση. Έχουμε φυσικά και κοινωνικές προκλήσεις. Ο τομέας των μεταφορών ε, απασχολείται και από το θέμα του κοινωνικού ντάμπινγκ και φυσικά εσείς είστε και η Φιλανδική Προεδρία, επομένως θα μας πείτε τα βασικά στοιχεία για την τεχνολογία ε, που ε, έχουμε προχωρήσει στην Ευρώπη, στα ψηφιακά ζητήματα. Θα μας πείτε λοιπόν αυτά τα νέα στοιχεία και το τελευταίο που είναι πολύ σημαντικό είναι να ακούσουμε κάποιες νέες ιδέες ε, για, να, ε, για που είναι πολύ σημαντικούς για μας, όπως ο τομέας της ναυτιλίας ε, και των αεροπορικών μεταφορών. Θα είμαι πάρα πολύ αυστηρή με το χρόνο στη διάρκεια της συζήτησης. Θα δώσω 10 λεπτά στην κάθε μία από εσά. Μετά θα γίνει ένας πρώτος γύρος με τους συντονιστές. Οι συντονιστές θα έχουν από δύο λεπτά ο καθένας για να θέσουν τις ερωτήσεις τους. Θα αφήσουμε χρόνο να απαντήσουν οι υπουργοί και από εκεί και πέρα θα υπάρχει ένας δεύτερος γύρος παρεμβάσεων. Καλώς ορίσατε λοιπόν στην Επιτροπή Μεταφορών. Κύρια Υπουργέ Μεταφορών, έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμότατα για τα ευγενικά σας λόγια. Χαίρομαι και εγώ ιδιαίτερος που είμαι εδώ μαζί σας σήμερα για να συζητήσουμε θέματα μεταφορών. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, νιώθω ιδιαίτερη χαρά που είμαι μαζί σας σήμερα για να εξετάσουμε και να συζητήσουμε τις προτεραιότητες του, της Φιλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου. Οι Ευρωπαίοι περιμένουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση θετικέ και συγκεκριμένε δράσει που θα επηρεάσουν την καθημερινότητά του. Για να υλοποιήσουμε αυτά τα αποτελέσματα, θα πρέπει να συνεργαστούμε στενά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει τεράστιε προκλήσει. Χρειαζόμαστε λοιπόν πρακτικά και ουσιαστικά μέτρα για να αντιμετωπίσουμε τόσο τι κλιματικέ αλλαγέ, αλλά και για να προετοιμαστούμε για αυτέ. Θα πρέπει επίση να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τι ευκαιρίε που μα δίνει ο ψηφιακό μετασχηματισμό. Η αλλαγή απαιτεί τόλμη, αφοσίωση και πάθος. Και το επίκεντρο όλων των δράσεών μας θα πρέπει να είναι ο πολίτης. Τι ρόλο λοιπόν θα διαδραματίσουμε. Θα χαράξουμε το δρόμο για νέες ιδέες, ε, δημιουργώντας πρόσφορο έδαφος για αλλαγές. Η βασική μας αρχή είναι να αντιμετωπίσουμε τις βασικές προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις και να τις εφαρμόζει κιόλα. Το σημαντικό είναι το αποτέλεσμα, το έργο, να παρουσιάσουμε έργο. Ε, Γενικώ, οι προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Προεδρία ε, ακολουθούν τα βασικά στοιχεία τη νέα στρατηγική ατζέντα, του νέου στρατηγικού θεματολογίου. Στόχο είναι να δημιουργήσουμε ε, ευζοία και ευμάρεια που θα είναι βιώσιμε κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά. Ο στόχος μας είναι μια ισχυρή, ενωμένη και εύρυθμα λειτουργούσα Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον τομέα των μεταφορών αντιμετωπίζουμε μείζωνα ζητήματα. Πώ να βελτιώσουμε τι υποδομέ, να μειώσουμε τι ε, εκπομπέ και να αξιοποιήσουμε πλήρω την ψηφιοποίηση και τι νέε τεχνολογίε. Σε ό,τι αφορά τι μεταφορέ, η Φιλανδική Προεδρία έχει εντοπίσει τέσσερι ε, στρατηγικού τομεί. Ψηφιακέ υπηρεσίε μεταφορών, αυτοματοποίηση τη μεταφορέ, ε, μεταφορέ απαλλαγμένε από τον άνθρακα και οικονομία των δεδομένων. Θεωρώ ότι αν επικεντρωθούμε σε αυτούς τους τομείς θα επιτρέψουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σημαντική και άμεση μείωση εκπομπών στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται και είναι απαραίτητη προπόθεση για να ελοπίσουμε του στόχου μα για τι κλιματικέ αλλαγέ. Τα δεδομένα και οι καλέ ιδέσει είναι βασικοί παράγοντε για να έχουμε απρόσκοπτε, αποδοτικέ οικονομικά και φιλοπεριβαλλοντικέ υπηρεσίε μεταφορών. Γι' αυτό και έχουμε επιλέξει το σύνθημα έξυπνε συνδέσει για βιώσιμη ανάπτυξη. Έτσι, ε, έχουμε το συνδυασμό των μεταφορών και των επικοινωνιών στην ψηφιακή εποχή και ε, αναφέρουμε και τις ε, ε, μελλοντικέ ανάγκες για την ανάπτυξη δικτύων. Θα πρέπει όλα αυτά να είναι με έξυπνο και βιώσιμο τρόπο. Αξιόπιστες υπηρεσίες μεταφορών που θα έχουν ως επίκεντρο τον πολίτη είναι η ραχοκοκαλιά μιας ανταγωνιστικής και εύρυθμα λειτουργούσας κοινωνίας. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε συνολικά την νομοθεσία και να δούμε τι μέσα μεταφοράς χρειαζόμαστε. Σίγουρα θέλουμε διαλειτουργικότητα και μια ευρύτερη κάλυψη και διαφορετική κάλυψη των υπηρεσιών μεταφοράς θα επιτρέψει τον, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Επίσης, ε, λύσεις αυτόματης και ασφαλούς ε, μεταφοράς θα πρέπει να προωθούνται. Η αυτοματοποίηση είναι βασικό στοιχείο για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά τι μεταφορέ, η αυτοματοποίηση θα συμβάλλει στην ε, βελτίωση τη ασφάλεια και τη αποτελεσματικότητα και στην επίλυση των κλιματικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων. Τα δεδομένα θα πρέπει να αποτελέσουν το βασικό καύσιμο για ένα βιώσιμο σύστημα ευρωπαϊκών μεταφορών. Θα πρέπει λοιπόν ε, να αξιοποιήσουμε τα, τα δεδομένα για να έχουμε αυτά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, τα αυτόματα οχήματα και η κινητικότητα ως υπηρεσία θα πρέπει να αναπτυχθούν με ταχύς ρυθμούς. Με τα δεδομένα θα επικεντρωθούμε καλύτερα στο χρήστη, θα έχουμε οικονομικά αποδοτικές και φιλοπεριβαλλοντικές υπηρεσίες μεταφορών και για να αναπτύξουμε τέτοιες ψηφιακές υπηρεσίες και αυτοματοποίηση θα πρέπει να αυξήσουμε και την πρόσβαση στα δεδομένα, την διαλειτουργικότητα των δεδομένων, αλλά να βελτιώσουμε και την ποιότητα και την επεξεργασία των δεδομένων. Με αυτά όλα κατά νου, το, ο στόχος της Φιλανδίας είναι να δώσει ενάψματα για την ε, πανευρωπαϊκή συζήτηση γύρω από τις αρχές της οικονομίας των δεδομένων. Ένα βασικό στοιχείο της ε, Προεδρίας μας και προτεραιότητάς μας είναι να πρωτοστατήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις κλιματικές δράσεις. Θέλουμε μια ε, ε οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, ανταγωνιστική χωρί κοινωνικού αποκλεισμού. Θα πρέπει επίση σε όλου του τρόπου, σε όλα τα μέσα μεταφορά, να μειώσουμε τι εκπομπές με οικονομικά αποδοτικό τρόπο και οι δυνατότητες που δίνουν η ψηφιοποίηση και η αυτομετοποίηση στη μείωση των εκπομπών θα πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως. Η μετάβαση από μια οικονομία με βάση τα ορυκτά καύσιμα σε μια οικονομία με χαμηλή χρήση άνθρακα έχει κέρια σημασία και είναι σημαντική και για μεταφορές όπως και σε άλλους κλάδους. Αυτό θα το ε, αναφέρουμε και θα το θέσουμε ως ζήτημα στο Συμβούλιο Μεταφορών του Σεπτεμβρίου. Η Φιλανδική Προεδρία ε, είναι προσιλωμένη στη συνέχιση του έργου για, τις, ε, για τους εκκρεμείς τομείς, για τις εκκρεμείς νομοθετικές πράξεις, δράσεις και στην περίπτωση των χερσαίων μεταφορών θα επικεντρωθούμε στα στα θέματα της Ευρωβινιέτας και των δικαιωμάτων των επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών προκειμένου να καταλήξουμε σε γενική προσέγγιση. Επίσης θα ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις για τον κοινωνικό πυλώνα και τον πυλώνα της αγοράς στο πρώτο πακέτο κινητικότητας όταν συμφωνήσετε στη συμφωνία. Θα συνεχίσουμε σε ό,τι αφορά τις, τα τέντη, τα διευρωπαϊκά δικτύα μεταφορών, τα θέματα δικτύων και διατροπικών ζητημάτων με στόχο να ξεκινήσουμε, να υλοποιήσουμε συμφωνία σε πρώτη ανάγκη ανάγνωση. Αν μα το επιτρέπει ο χρόνο, θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε και διαπραγματεύσουμε το Κοινοβούλιο. Σε ό,τι αφορά το ηλεκτρονικό σύστημα για τι ε, μεταφορές, τις ηλεκτρονικέ εμπορευματικέ μεταφορέ, επίση θα συνεχίσουμε τι ε, συζητήσει, καθώ και για το θέμα τη θερινή ώρα. Σε ό,τι αφορά την ε, αεροπορία, θα συνεχίσουμε τι διαπραγματεύσει με τρίτε χώρε για να συνάψουμε συμφωνίε και να επαναφέρουμε στην συζήτηση το θέμα των δικαιωμάτων των επιβατών αερομεταφορών. Θα πρέπει όμω πρώτα το Συμβούλιο να κάνει ένα απολογισμό τη παρούσα κατάσταση, γιατί η τελευταία φορά που συζητήσαμε την πρόταση στο Συμβούλιο ήταν πριν από μία τετραετία. Στην αυτιλία επίση. Θα συντονίσουμε τις θέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας. Επιπλέον θα φροντίσουμε και θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε τον παγκόσμιο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα βιωσιμότητα, ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση. Στη διάρκεια τη προεδρία μα, θα οργανώσουμε πολλέ εκδηλώσει για να δώσουμε ενάσματα για τη συζήτηση για το μέλλον των μεταφορών και τη πολιτική επικοινωνία. Επ' ευκαιρία θα ήθελα να σα ενθαρρύνω και να σα καλέσω όλου να συμμετέχετε σε αυτό το διάλογο. Θα οργανώσουμε διασκέψει ενδιαφερομένων μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι ημερίδε ψηφιακών μεταφορών θα προσφέρουν το, ευρωπαϊκό τρόπο σκέψης για ψηφιακές λύσεις στην κινητικότητα και τις μεταφορές. Θα πρέπει να συμβάλλουμε να δημιουργηθεί μια ε, όθηση για να συζητήσουμε και το θέμα των ενιαίων ευρωπαϊκών εθέρων στη διάσκεψη ψηλού επίπεδου για το μέλλον του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού. Ε, η διάσκεψη ψηλού επίπεδου για την οικονομία των δεδομένων θα οργανωθεί προκειμένου να διερευνήσουμε το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας των δεδομένων. Δύο συμβούλια μεταφορών θα έχουμε στη διάρκεια τη Φιλανδική Προεδρία. Στι 20 Σεπτεμβρίου θα έχουμε συμβούλιο μεταφορών στι Βρυξέλλες, προκειμένου να εξετάσουμε ε, τις, ε, τα θέματα της μεταφοράς ό,τι αφορά το στρατηγικό μακροπρόθεσμο στόχο και όραμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση για μια ε, οικονομία που θα είναι ουδέτερη για το κλίμα. Και το δεύτερο Συμβούλιο Μεταφορών θα γίνει στι 2 ή 3 Δεκεμβρίου του 2019 στις Βρυξέλλες, αν θυμάμαι καλά. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτέ, τα θέματα των μεταφορών απασχολούν διαρκώς την κοινή γνώμη και μας δίνουν ξεκάθαρες ενδείξεις για το πώς ε, η πολιτική μεταφορών επηρεάζει την καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών. Και οι πολίτες και ο κλάδος περιμένουν πολλά από μας. Ε, ο πύχης έχει μπει πολύ ψηλά και αυτό θα μας παροτρύνει να εργαστούμε πιο αποτελεσματικά και να λάβουμε αποφασιστικές δράσεις για να υλοποιήσουμε τους κοινού μας στόχους. Και μια ε, και διαπιστώσετε από το μακροσκελή κατάλογο ότι έχουμε πολλά θέματα μπροστά μας. Ε, θα, σας, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω για την προθυμία μου να εγγύψουμε με ενθουσιασμό σε αυτό το έργο και η συνεργασία μας θα, διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για να προωθήσουμε τα θέματα αυτά και να σημειώσουμε πρόοδο. Με ενδιαφέρει λοιπόν να δω πώς θα συνεργαστούμε Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να αντιμετωπίσουμε από κοινού τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Όπως είπα και στην αρχή, θεωρώ ότι η πρωταρχική και μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ψηφιοποιήσουμε τον τομέα των μεταφορών και να το καταστήσουμε ουδέτερο από την άποψη του άνθρακα και των ανθρακούχων εκπομπών. Σας ευχαριστώ. Κίτος που λέμε και στα φιλανδικά. Vous voyez, quand on dit 10 minutes, c'est 10 minutes. Bravo. Μπράβο σας, είπα 10 λεπτά, το τηρήσατε πιστά. Βλέπετε ότι είναι υπερφορτωμένη η μερίσια διάταξη ε, και για το, Υπουργείο, το Συμβούλιο Μεταφορών και είπατε μια πολύ σημαντική φράση. Ήρθε η ώρα να περάσουμε σε αλλαγέ. Ε, πέρασε ε, ο καιρός για τα λόγια, θα πρέπει να περάσουμε στα έργα, στις πράξεις. Και φαίνεται ότι όλοι είμαστε έτοιμοι, ενθουσιασμένοι να ανασκουμποθούμε και να περάσουμε στα έργα. Και ένα μείζον ζήτημα που επισημάνετε κι εσείς είναι το θέμα των κλιματικών αλλαγών. Και τώρα θα δώσω το λόγο στη συνάδελφό σας, ε, την Υπουργό Τουρισμού. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί Ευρωβουλευτές, είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά που βρίσκομαι εδώ πέρα σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελπίζω να βλεπόμαστε συχνά κατά τη διάρκεια της Φιλανδικής Προεδρίας και μετά. Και αναμένω βεβαίω την ένταση της συνεργασίας μας για την Ευρωπαϊκή Προεδρία. Χαίρομαι που έχω αυτή την ευκαιρία σήμερα να συζητήσω μαζί σας την Φιλανδική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Φιλανδία έχει έναν φιλόδοξο στόχο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει η πιο ανταγωνιστική οικονομία και ταυτόχρονα να είναι ουδέτερη ως προς το κλίμα. Ελπίζουμε λοιπόν να πετύχουμε αυτόν το, αυτό το κοινό μας όραμα για μια νέα ατζέντα για την ανάπτυξη. Η Προεδρία μας θεωρεί ότι τα βασικά στοιχεία θα περιλαμβάνουν την μετάβαση προς μια οικονομία ουδέτερη ω προς το κλίμα, αποτελεσματική ενιαία αγορά, σύγχρονη βιομηχανική πολιτική με ψηφιακή οικονομία, καινοτομία, ενεργή εμπορική πολιτική και νέες ε, δεξιότητες. Οι κοινέ μας ε, προσπάθειες χρειάζονται έτσι ώστε οι στόχοι αυτοί να γίνουν πραγματικότητα. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, με χαρά σας μιλάω σήμερα για τον ε, τουρισμό. Έναν βασικό στρατηγικό κλάδο με πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες για την ανάπτυξη. Ο τουρισμός εξακολουθεί να έχει μια όλο ένα αυξανόμενη σημασία για την οικονομική ανάπτυξη, περιφερειακή ανάπτυξη για την απασχόληση. Είναι πάνω από 10% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ και σχεδόν 12% των εργαζομένων εργάζονται στον ε, τουρισμό. Μετά την επιτυχημένη Ρουμανική Προεδρία και η Φιλανδία θα συνεχίσει την συζήτηση στο θέμα της πολιτικής του τουρισμού. Κατά τη διάρκεια της Ρουμανικής Προεδρίας, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου ανέδειξαν την ανταγωνιστικότητα στον τομέα του τουρισμού ως ένα θέμα το οποίο θα μπορούσε να προσφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη, τις δουλειές, την κοινωνική συνοχή, την αηφόρο καινοτομία και την ψηφιοποίηση αποτελεί βεβαίως ε, παράγοντες επιτυχίας αλλά και προκλήσεις. Η κύρια προτεραιότητά μας είναι να δώσουμε συνέχεια στα συμπεράσματα αυτά και να προωθήσουμε την ψηφιοποίηση του τομέα του τουρισμού. Χρειάζεται συζήτηση για τα επόμενα βήματα για να προωθήσουμε την πολιτική τουρισμού περαιτέρω στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αγαπητοί η ψηφιοποίηση είναι στρατηγικό τομέα συνεργασία για να επιταχυνθεί η ανάπτυξη, η ευημερία και η απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται πολιτικέ τουρισμού οι οποίε θα μπορέσουν να δουν το θέμα τη γρήγορη εξέλιξη τη ψηφιοποίηση. Τα καθήκοντα τη νέα ε, Κομισιόν αλλά και των κρατών μελών είναι να δούμε πώ θα μπορέσουμε να μεγιστοποιήσουμε τι ευκαιρίε ε, και την ανάπτυξη της ψηφιοποίηση στον τομέα του τουρισμού για τις επιχειρήσεις, ε, τους ε, ταξιδιώτες και τις τοπικές ε, κοινωνίες. Το βασικό ερώτημα είναι το εξής. Ποια μέτρα πρέπει να λάβουν τα κράτη-μέλη και η Κομισιόν για να διασφαλιστεί ότι ο τομέας του τουρισμού θα επιτύχει στη μαγκοσμία οικονομία. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, θα ήθελα να σα παρουσιάσω τρει τομεί κλειδιά τη ψηφιοποίηση στον τομέα τουρισμού. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να υπάρχει καλύτερη διαχείριση δεδομένων στον τομέα τουρισμού. Δεύτερον, η παρουσία του τομέα τουρισμού στα ψηφιακά δίκτυα πρέπει να αυξηθεί. Πρέπει να υπάρχει καινοτομία. Τρίτον, χρειάζεται να αναπτυχθούν ψηφιακές δεξιότητες ε, στις τουριστικές επιχειρήσεις, ειδικά τις μικρομεσαίες. Συνοψίζοντας, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, χρειάζεται οικονομική ανάπτυξη και πρέπει να είναι βιώσιμη περιβαλλοντικά και κοινωνικά. Ένα νέο σχεδιασμό για την ανάπτυξη είναι απαραίτητος ε, για να πάμε προς μια κοινωνία ουδέτερη ω προς το κλίμα. Α θέσουμε μαζί αυτόν τον ε, στόχο λοιπόν. Πρέπει να προωθήσουμε μια ανταγωνιστική ένωση η οποία θα περιλαμβάνει τους πάντες και θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών της. Αναμένω λοιπόν την συζήτηση μαζί σας και την ανταλλαγή απόψεων για την τουριστική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Υπουργέ. Στην Επιτροπή αυτή ο τουρισμός ε, είναι ένας ε, τομέας προτεραιότητας ε, και όπως είπαμε στη συνεδρίαση των συντονιστών θα ενισχύσουμε αυτή την ψυχή για να μπορέσουμε κάτι καλύτερο για το αύριο. Και έχετε δίκιο. Ε, χρειαζόμαστε κάτι βιώσιμο, αποδεκτό και κυρίως προσβάσιμο. Και επομένως ε, τώρα θα ξεκινήσει η συζήτηση και θα ξεκινήσω με τους συντονιστές. Ο κύριος Μαρινέσκου από το ΕΛΚ δεν είναι εδώ, δεν ξέρω ποιος ε, θα τον αντικαταστήσει. Η κυρία Τέντερ, για δύο λεπτά. Παρακαλώ να είστε σαφείς, συγκεκριμένοι. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητές Υπουργέ, σας ευχαριστώ για την παρουσίαση και για τα φιλόδοξα σχέδια για τις μεταφορές και για τον τουρισμό. Η Ευρωβινιέτα είναι πολύ σημαντικό θέμα για μας. Η ευρωπαϊκή οικονομία, καθώς και η εθνική μας οικονομία ε, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό σε προσβάσιμες και αποδοτικές μεταφορές για να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Και επίσης ε, πρέπει να διατηρήσουμε και την κοινωτικότητα των πολιτών και το δικαίωμα να επιλέγουν το μέσο μεταφοράς που επιθυμούν. Τι θα κάνετε με τα περιβαλλοντικά ζητήματα και τα θέματα επικουρικότητας από την άλλη. Τι μπορούμε να περιμένουμε από την γενική προσέγγιση. Τώρα, ο ενίος Ευρωπαϊκός Ουρανός. Εμείς ως ΕΛΚ ε, θέλουμε να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό και να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Αν υπάρχει προθυμία από πλευρά Συμβουλίου, θα μπορούσε να είναι τεράστιο επίτευγμα αυτό για την Ευρώπη. Το περιβάλλον και φυσικά και για τη Φιλανδική Προεδρία. Ο συνάδελφος Άντορ Ντέλη θα ερω... Ε, θέσει ερωτήσεις ε, για το πακέτο των μεταφορών σε συνέχεια, αλλά εμείς ως ΕΛΚ, όπως και άλλες πολιτικές ομάδες, ε, είμαστε διαιρημένοι για τη δέσμη αυτή. Δύο λόγια τώρα για την ψηφιοποίηση. Εδώ και 12 χρόνια εγώ είμαι επιχειρηματία στο τομέα της πληροφορικής, επομένως διαφάζω πολύ προσεκτικά τα σχέδια και το πρόγραμμά σας για την ψηφιοποίηση το, του τομέα των μεταφορών. Θα μπορούσατε ίσως να μας πείτε κάποιες λεπτομέρειες επιπλέον και θα μπορούσα να, να μας πείτε και ένα-δυο πρωτοβουλίε ε, ε, πέραν του ΙΦΡΕ που θέλετε να αντιμετωπίσετε στις, ε, στην Προεδρία σας. Τώρα θα μιλήσω γερμανικά για την τελευταία ερώτηση. Οι συγκοινωνίες ε, και ο τουρισμός υπάρχουν ήδη στις συνθήκες της ε, Ρώμης. Ε, αποτελούν βασικό κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά υπάρχουν και κάποιες σκοτεινές πτυχές. Εγώ επειδή είμαι από το Τυρόλο αναρωτιέμαι τι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να επιτύχει τον στόχο της μείωσης των βαρέων οχημάτων κατά 30% μέχρι το 2030, ειδικά στην περιοχή της, ε, του Μπρένερ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ερτούγ από τους Σοσιαλιστές. Ναι, καλημέρα σε όλους και όλες και πάλι. Καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και νομίζω πως ε, και οι δύο Υπουργοί Μεταφορών και Οικονομίας δείχνουν ότι στους ε, τομείς αυτούς ε, βιομηχανίας, μεταφορών, κινητικότητας και περιβάλλοντος ε, πρέπει να τους δούμε από κοινού. Σας ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις σας. Έχω δύο-τρεις ερωτήσεις. Είναι προφανές ότι η Φιλανδία έχει κάποια εμπειρία σε αυτήν την οικονομία των δεδομένων λέτε κινητικότητα ως υπηρεσία, ψηφιακές υπηρεσίες. Ο κλάδος ε, συζητάει τόσα πράγματα για τα νέα αυτά μοντέλα. Θα ήθελα να ακούσω κάποια πράγματα για τις εμπειρίες σας στη Φιλανδία. Συγκεκριμένα για τις έξυπνες συνδέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη, νομίζω έτσι το είπατε. Μπορείτε να μας δώσετε κάποια παραδείγματα από τη Φιλανδία, τι έχετε ήδη κάνει και ποιος ήταν ο αντίκτυπος, ήταν ε, επιτυχημένη προσπάθεια, όχι, εύκολη, δύσκολη. Αυτό θα έχει μεγάλη σημασία νομίζω για την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρώτη ερώτηση είναι αυτή. Η δεύτερη. Θέσατε το ζήτημα της ανάπτυξης των αυτόνομων οχημάτων. Έχετε κάποιες ε, περιφέρειες όπου δοκιμάζετε αυτά τα μέσα. Και τρίτον, μιλήσατε για τα εκρεμή ζητήματα, συγκεκριμένα τα δικαιώματα επιβατών σιδηροδρόμων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία. Αναφέρατε την Ευρωβινιέτα και οπωσδήποτε το πακέτο κινητικότητας 1 ε, δεν με ενδιαφέρει πολύ αυτό. Νομίζω πως η Προεδρία οπωσδήποτε έχει δεσμευτεί να το προχωρήσει. Θα ήθελα να γνωρίζω κάποια πράγματα περισσότερα για τους σιδηρόδρομους. Έχετε κάποιες ιδέες ως Προεδρία για το ζήτημα αυτό. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ακριβώς για να μπορέσουν να ακολουθήσουν και τα κρατη Αυτά, αυτά για την ώρα. Σας ευχαριστώ και πάλι. Σας, Σας ευχαριστώ κύριε Έρτουγκ. Η κυρία Νάστιγκαλ. Α, εσείς θα μιλήσετε τελικά. Ο κύριος ε, Μπόζας. Σας ευχαριστώ. Θα Φεύγω γιατί έχω ένα ραντεβού με κάποιον υπουργό. Δίνω το λόγο στον συνάδελφο. Απλώ αυτό ήθελα να πω. Η κυρία Σντεγκάλ έχει το λόγο. Ευχαριστώ που ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι δυο σα. Και μα δίνετε και την ευκαιρία να σα θέσουμε κάποιε ερωτήσει για την Φιλανδική Προεδρία του Συμβουλίου. Δύο σύντομε ερωτήσει η οποία αφορά και τη νέα εντολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις νέες ε, πολιτικές ομάδες και εμείς ως νέα πολιτική ομάδα είμαστε πλέον το Renew Europe και θα θέλαμε να κάνουμε τα πράγματα διαφορετικά για να μπορέσουμε πραγματικά να ανανεώσουμε την Ευρώπη. Πώς ε, θα τιμήσει την ονομασία μας λοιπόν η Φιλανδική Προεδρία, τι θα κάνατε λοιπόν για να ε, δείξετε ότι κάνετε κάτι διαφορετικό από τις προηγούμενες προεδρίες. Η δεύτερη ερώτησή μου ως Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε κατά νου τα συμφέροντα όλων των χωρών. Ωστόσο, διαπιστώνουμε κάποιες φορές ότι υπάρχουν κάποιες διαφορές ε, στα συμφέροντα μεταξύ ε, νότου, βορρά, ανατολικών και δυτικών ε, χωρών. Πώς θα μπορέσει ειλικρινά να μεσολαβήσει η Προεδρία σας μεταξύ των διαφορών χωρών. Ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος των Πρασίνων, η κυρία... Α, συγγνώμη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και καλωσορίσατε να πω στις υπουργού. Είναι τιμή να σας έχουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η πρώτη με ερώτηση απευθύνεται στην Υπουργό Τουρισμού. Γνωρίζουμε ότι η οικονομική και περιβαλλοντική αξία του ποδηλατικού τουρισμού είναι ανεκτήμητη πάνω από 2 δισεκατομμύρια ε, ετήσιοι γύρι με αξία ε, πάνω από 4 δις ευρώ. Και αυτό σχετίστηκε με πάνω από 2.000 θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι σκοπεύετε να κάνετε λοιπόν εσείς στην Προεδρία σας για να δώσετε όθηση σε τέτοια περιβαλλοντικό, βιώσιμο και οικονομικά πάρα πολύ σημαντικό τύπο τουρισμού. Η δεύτερη ερώτηση είναι προς την Υπουργό Μεταφορών. Γνωρίζουμε βεβαίως ότι όταν αναφερόμαστε στην κινητικότητα ως υπηρεσία, ε, τα μέσα μαζικής μεταφοράς ε, και η ενεργός κινητικότητα θα πρέπει να είναι βασικοί πυλώνες. Όσον αφορά την αυτοματοποίηση, πώς λαμβάνετε υπόψη ε, το κίνδυνο της ατομικής κινητικότητας, όπως περνάμε στην αυτοματοποίηση, μπορεί να μειωθεί το ποσοστό ε, κατοχής αυτοκινήτων και να αυξηθεί η κίνηση. Βλέπουμε, έχουμε δει όλοι ε, ο καρτούν με την εικόνα της κίνησης σήμερα και της κίνησης όταν θα είναι αυτοματοποιημένη και δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ των δύο στην κυκλοφοριακή συμφόρηση. Τι θα κάνετε εσείς ώστε να μειωθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση όσο προχωρούμε σε μεγαλύτερη αυτοματοποίηση. Και μια δεύτερη ερώτηση για τις μεταφορές, για τις αεροπορικές μεταφορές. Πολλοί από εμά υποστηρίζουν ε, τη μεταφορά ε, σε σημαντική φορολόγηση της κυροζήνης για τις αεροπορικές μεταφορές και θα ήθελα να ξέρω τι σκοπεύετε να κάνετε εσείς ε, στη διάρκεια της Προεδρίας σας για να προωθήσετε αυτή την πρόταση. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε, κύριε Κόφ. Περνάμε στην ομάδα ID, Ταυτότητα και Δημοκρατία, που είναι ο συντονιστής. Ο κύριος Καμπονάζο. Ναι, το επίθετό μου είναι λίγο δύσκολο, αλλά θα το μάθετε, θα το προφέρετε σιγά σιγά. Υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις που θα μπορούσα να κάνω. Καταρχάς, ε, και εγώ να σας καλωσορίσω με τη σειρά μου. Είναι ιδιαίτερη περίοδος αυτή που αναλαμβάνεται καθήκοντα, διότι έχουμε ένα σώμα επιτρόπων που σύντομα θα αποχωρήσει και θα έρθει ένα νέο σώμα επιτρόπων. Επομένως, οι σχέσεις με τον μελλοντικό επίτροπο μεταφορών θα είναι πολύ σημαντικό. Σήμερα θα δούμε και την ε, ε, παρούσα επίτροπο, την κυρία Μπουσκόλοι βέβαια ενδιαφέρονται ε, να μάθουν τι θα γίνει με το πακέτο για την κινητικότητα. Στην προηγούμενη θητεία η ομάδα μου ε, ήταν αναφανδόν υπέρ ε, των θεμάτων και η κυβέρνηση της χώρας μου είναι υπέρ και γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχουν δυσκολίες παρόλα αυτά. Όπω ε, και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, θα ήθελα να γνωρίζω τι θα μπορούσατε να κάνετε προκειμένου να προσπαθήσετε να διευκολύνετε ε, την εξέβρεση λύση που θα βοηθήσει και τι χώρε τη Ανατολική Ευρώπη, που σήμερα είναι αυτέ που διαμαρτύρονται. Αλλά πιστεύω ότι συνειδητοποιούν και αυτέ ότι οι χώρε τη Δύση έχουν και αυτέ ε, την ανάγκη να καταπολεμήσουν κάποιες αθέμητε πρακτικέ και έναν ανταγωνισμό ο οποίο δίνει κίνητρα για ψευδή μεταφορά επιχειρήσεων Προ τι ανατολικέ χώρε, ε, οι οποίε ε, υποτίθεται ότι δραστηριοποιούνται στι ανατολικέ χώρε, αλλά τελικά χάρη στην εσωτερική αγορά δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στη Γαλλία, στην Ιταλία, στη Γερμανία και στην Αυστρία και όχι μόνον. Όσον αφορά τι αεροπορικέ μεταφορέ, θα θέλαμε να υπάρξει κάποια πρόοδο. Ε, θα θέλαμε να ξέρουμε αν έχετε κάποιες ιδέε για τον ενιαίο ουρανό, ώστε να μπορέσει να ξεμπλοκάρει και ένα πολύ λεπτό θέμα που αφορά το Γιβραλτάρ. Και όλοι ξέρουμε ότι βρίσκεται στο επίκεντρο του προβλήματος αυτού. Ε, θα θέλαμε να ξέρουμε λοιπόν αν υπάρχει κάποια στρατηγική επ' αυτού που να συνδέεται ίσως και με το Brexit, ε, που θα μπορούσε ίσως να περιπλέξει, αλλά και να απλοποιήσει τα πράγματα. Δεν ξέρω, θα το δούμε όλοι μαζί κάποια στιγμή. Κάποιος πριν από μένα αναφέρθηκε στον Μπρένερο στην Ιταλία ε, και τη Γερμανία, που πρέπει να βρουν ένα σημείο ε, συνάντησης στο θυμίο αυτό. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ να τηρείτε το χρόνο αγόρευσης. Είπα ένα λεπτό, αλλιώς θα σας ε, παίρνω το μικρόφωνο. Και το ένα λεπτό ισχύει για όλους. Παρακαλώ, συνάδελφε Λεμπρεζέ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλωσορίζω και τις δύο υπουργέ στην Επιτροπή Μεταφορών. Τις δύο υπουργούς, συγγνώμη. ευχαριστώ για την παρουσίαση. Εγώ θα ξεκινήσω με το πρώτο πακέτο κινητικότητας που αναφέρθηκε από κάποιους Είπατε ότι περιμένετε την εντολή και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την έναρξη των διαπραγματεύσεων και ξέρετε ότι μερικοί υπουργοί μεταφορών βρίσκονται ήδη σήμερα στις Βρυξέλλες αλλά η κατάσταση είναι ακόμη ασαφής. Δεν ξέρουμε ποιοι κανόνες ισχύουν ε, για την διαμόρφωση θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με τη θέση που έχει προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία. Θα πρέπει να γίνουν κάποια συγκεκριμένα βήματα λοιπόν να θέλουμε να αρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις για το πρώτο πακέτο κινητικότητας. Είναι σαφές ότι υπάρχει διχόνοια μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Ευρωπαϊκών χωρών διάσταση απόψεων για το πακέτο κινητικότητας. Σε ό,τι αφορά τις, ε, τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου αν εγκριθούν οι παρούσες ε, διατάξεις για τη μεταφορά των φορτηγών, δεν θα έχουμε πραγματικές ε, μειώσεις εκπομπών ε, που θα είναι και οικονομικά αποδοτικές. Επίσης είπατε για, την, για το άνοιγμα των αγορών που επιτρέπεται κυρίως από το δεύτερο πακέτο κινητικότητας. Υπάρχει κάποια προθυμία από το Συμβούλιο για να προχωρήσουμε στο μέλλον με αυτό το θέμα, το δεύτερο πακέτο κινητικότητας. Ε, για το συνδέοντα στην Ευρώπη θα μιλήσετε με τους Υπουργούς Μεταφορών. Γιατί υπήρχε κάποια αντίφαση με την αρχική θέση της Ευρω... μεταξύ της αρχικής θέσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κοινοβουλίου με το πώς θα συνδυάσουμε το συνδέοντα στην Ευρώπη, το Ταμείο Συνοχής και τα μεγαλεπίβολα σχέδια μεταφορών στην Ευρώπη. Ευχαριστώ κύριε Κουντουρά για δύο λεπτά. Εκ μέρους της ΓΚΟΕ. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω για τις ε, εισαγωγικές σας παρατηρήσεις, ε, κυρία Υπουργοί, και να σας ευχηθώ μια επιτυχημένη Προεδρία του Συμβουλίου. Διάβασα το πρόγραμμά σα, εντόπισα δύο βασικού πυλώνε, όπω και εσεί αναφερθήκατε, για την ψηφιοποίηση και τη μείωση των ρήπων, οροματική και μακροπρόθεσμη στόχη. Θα ήθελα λοιπόν να σα ρωτήσω πώ θα κινηθείτε, ποια συγκεκριμένα βήματα θα κάνετε στην εξάμηνη προεδρία σα για να προχωρήσετε στου στόχου αυτού, λαμβάνοντα υπόψη ότι και τα 27 κράτη-μέλη έχουν διαφορετικά σημεία κίνηση. Θα ήθελα επίσης, να, και εγώ από τη μεριά μου, να σας καλέσω να θέσετε ως βασική προτεραιότητα τη Προεδρία σα και να δεσμευτείτε ότι θα καταβάλλετε κάθε προσπάθεια να βρεθεί μια συμφωνία στο πακέτο κινητικότητας που θα σέβεται τις βασικές θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διότι πρέπει να σημειώσουμε ότι θα βελτιώσει σημαντικά τα δικαιώματα των εργαζομένων στο κλάδο αλλά και θα συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της ασφάλειας στους ευρωπαϊκούς αυτοκινητόδρομους. Στον τουρισμό θα ήθελα να πω ότι επειδή υπήρξα και εγώ υπουργό τουρισμού και γνωρίζω ότι η βιώσιμη ανάπτυξη είναι και υπεύθυνη ανάπτυξη και ο κλάδος των μεταφορών συνδέεται με τον τουρισμό αλλά και αντίστροφα, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν σκοπεύετε να στηρίξετε την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη δημιουργία ενός σοβαρού προϋπολογισμού για τον τουρισμό στο επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και αν σκοπεύετε να επανεκκινήσετε τις εργασίες για μια στρατηγική ώστε η Ευρώπη να έχει μια ενιαία τουριστική πολιτική και να παραμείνει κορυφαίος τουριστικός παγκόσμιος προορισμός. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Νομίζω ότι θα χρειαζόταν μία ώρα μία για να απαντήσετε, αλλά δυστυχώ δεν έχουμε τόσο χρόνο. Λίγα λεπτά μόνο, αλλά ευτυχώ μερικέ ερωτήσει επαναλαμβάνονται. Το θέμα του πρώτου πακέτου κινητικότητα των δικαιωμάτων των επιβατών. Και θα ήθελα να υπογραμμίσω το θέμα των δικαιωμάτων επιβατών, γιατί όταν λέμε 8 θέσει σε όλα τα τρένα, εννοούμε 8. Οπότε και κοιτάω εδώ τον κύριο Λιμπεράτσκι που είναι ο αρμόδιος ε, για τα θέματα αυτά, ενώ συγκεκριτή μας, θα ήθελα να τονίσω εδώ ότι είμαστε ανένδοτοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα δικαιώματα των επιβατών. Και το τονίζω αυτό. Και όταν λέμε 8 θέσεις ε, στα τρένα, είναι 8, ούτε 2 ούτε 3. Και το συνδέσαμε και με τον τουρισμό, με ε, τον ποδηλατικό τουρισμό. Επίσης, για τις φορές των φορτηγών, των τριαξονικών. Επίση, ε, το θέμα της αυτόνομης, αυτοματοποιημένη οδήγησης, ένα θέμα που επανήλθε σε πολλέ ερωτήσει και η οικονομία των δεδομένων. Όλα αυτά μα ενδιαφέρουν. Εσεί ε, πώ θα τα λάβετε υπόψη όλα αυτά στο πρόγραμμά σα, ε, αν έχετε εμπειρίε ήδη, τι προτάσει έχετε. Επίση, αεροπορία, ενιαίος ευρωπαϊκό ουρανό. Τι γίνεται, θα βάλετε όντω την ταχύτητα για να κινηθούμε γρήγορα σε όλα αυτά τα θέματα και ο τουρισμός επίσης είναι βασική αρμοδιότητα και της δικής μας Επιτροπής και σημαντικός κλάδος της Ευρωπαϊκής Οικονομίας. Θα δώσω πρώτα το λόγο στην Υπουργό Μεταφορών και κατόπιν στην αρμόδια Υπουργό για τον Τουρισμό. Στα φιλανδικά τώρα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους συντονιστές για τις πολύ εύστοχες ερωτήσεις τους και τις ε, αξιόλογες παρεμβάσεις τους. Κυρία Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο καλύτερα γίνεται σε αυτές τις ε, σημαντικές ερωτήσεις. Ε, τώρα τα θέματα τα φιλανδικά θα μπορούσα να τα αναφέρω, αλλά είναι μάλλον αντικείμενο άλλη συζήτηση. Πάντω, σα διαβεβαιώ ότι εμεί, ω Φιλανδική Προεδρία, θα εκπροσωπούμε το σύνολο του Συμβουλίου και όχι μόνο τα φιλανδικά θέματα. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσει η Φιλανδική Προεδρία να κρατήσει μια ουδετερότητα, μια μεροληψία, ακούγοντας όλους τους συνομιλητέ. Αυτό είναι σημαντικό μας μέλημα. Και στο πρώτο πακέτο κινητικότητας αναζητήσαμε συμβαστικέ λύσεις προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι διστάμενε απόψεις. Και έτσι θα συνεχίσουμε και στο μέλλον, με ουδετερότητα και ακούγοντα όλους του συνομιλητέ. Στι εισαγωγικέ μου παρατηρήσει σα μίλησα για τι βασικέ μα προτεραιότητε. Το θέμα των κλιματικών αλλαγών, για παράδειγμα. Και το πώ ε, ε, θα μειώσουμε τους ρήπους στις μεταφορές. Επίσης, ε, για το πρώτο πακέτο κινητικότητας, ο κοινωνικός πυλώνας και ο πυλώνας της αγοράς ήταν ακαθόδη ζητήματα στο Συμβούλιο. Σίγουρα δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό το πακέτο κινητικότητα υπαριθμών 1. Θα πρέπει να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ των κοινωνικών δικαιωμάτων των οδηγών αλλά και τη ε, παροχή υπηρεσιών σε μια ελεύθερη ανταγωνιστική αγορά. Και θέλουμε πιο αποτελεσματικέ υπηρεσίε. Και τον περασμένο Δεκέμβριο δεχτήκαμε στο Συμβούλιο Μεταφορών το πακέτο και περιμένει το Συμβούλιο την έναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αν γίνεται και στη διάρκεια της Φιλανδικής Προεδρίας. Εμείς είμαστε σε ετοιμότητα και ως έντιμοι διαμεσολαβητές θα αναζητήσουμε συμβαστικές λύσεις και επικοδομητικές με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαι πεπισμένη ότι θα έχουμε αγαστή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρόλο που τα ζητήματα αυτά είναι αρκετά δύσκολα. Σε ό,τι αφορά τις μεταφορές και την Ευρωβινιέτα, αυτό το θέμα το συζήτησε το Συμβούλιο τον Ιούνιο. Εκεί εξετάσαμε μια μελέτη πρόδου και επαναλαμβάνω, οι διαπραγματεύσει στο Συμβούλιο θα συνεχιστούν στη διάρκεια της Φιλανδικής Προεδρίας και θα προσπαθήσουμε να τις προχωρήσουμε όσο γίνεται. Θέλουμε να βρούμε ισορροπία μεταξύ της επικουρικότητας αφενός και των κλιματικών και περιβαλλοντικών πτυχών αφετέρου. Δεν μπορώ τώρα να πιθανολογήσω την τελική έκβαση των συζητήσεων. Είχαμε διμερεί συζητήσει με όλα τα κρατη Θα συνεχίσουμε τι διαπραγματεύσει στο Συμβούλιο το Σεπτέμβριο και γνωρίζω τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ευρωβινιέτα που είναι αποκρισταλωμένη. Σε ό,τι αφορά τι κλιματικέ δράσει για τον τομέα των μεταφορών, στόχο μα είναι να πρωτοστατήσει και παγκοσμίω η Ευρωπαϊκή Ένωση στα θέματα αυτά των κλιματικών αλλαγών. Ήδη δηλώσαμε την προσήλωσή μας στους στόχους των Παρισίων και Θέλουμε να στείλουμε στις αρχές του 2020 τους ε, στόχους μας. Τα περισσότερα κράτη-μέλη συμφώνησαν ε, να, έχουμε δράσει ουδέτερες ως προς το κλίμα μέχρι το 2050 και θέλουμε να βρούμε μια κοινή θέση. Το Συμβούλιο θα συνεχίσει τις συζητήσεις ε, και τα συμπεράσματά του θα αποτελέσουν τη βάση για τις αποφάσεις σας σε υψηλό επίπεδο. Και σίγουρα θα πρέπει να δώσουμε κάποια ενάψματα, κάποια κίνητρα για να διευκολύνουμε ε, την, ε, ένα κλάδο μεταφορών που θα είναι ουδέτερος κλιματικά. Όπως σας είπα, στις 20 Σεπτεμβρίου θα γίνει το πρώτο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών και θα επικεντρωθεί κυρίως στις κλιματικές προκλήσεις. Τέθηκε μία ερώτηση για τις υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες στηρίζονται συχνά στη χρήση ψηφιακών πληροφοριών, πολυτροπικότητα, χρήση νέων τεχνολογιών. Έχουμε τα ηλεκτρονικά πατίνια σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις πια. Έχουμε λοιπόν νέες υπηρεσίες που αξιοποιούν τις ψηφιακές ε, υπηρεσίες και θέλουμε να εξυπηρετούν τους Ευρωπαίους πολίτες. Με ρωτήσατε και για την αεροπορία και εκεί θέλουμε φιλόδοξες αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και παγκοσμίω προκειμένου να τηρηθεί η Συμφωνία των Παρισίων. Και πιστεύω ότι θα λάβουμε σημαντικές αποφάσεις στον τομέα αυτό. Και η αποτελεσματικότητα επίσης είναι σημαντικό θέμα και θα πρέπει να το δούμε και στην ΕΚΑΟ, στη Διεθνή Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας. Και το θέμα εμπορίας εκπομπών, το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Θα πρέπει να λαμβάνονται αποτελεσματικές αποφάσεις χωρίς να υπάρχει στρέβλωση του, εθνικού, του ανταγωνισμού σε εθνικό επίπεδο, χωρίς να υπάρχει αύξηση της γραφειοκρατίας και επίση να προωθήσουμε τη χρήση βιοκαυσίμων και στι αερομεταφορέ. Να βρούμε λοιπόν τρόπους ε, και να δώσουμε ενάμσματα στις αεροπορικές εταιρείες ε, για να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες. Τέθηκε μια ερώτηση για τις νομοθετικές προτάσεις για τις αερομεταφορές. Το 2013 η Ευρωπαϊκή Πρόταση υπέβαλε την Επιτροπή για τους ενιαίους ευρωπαϊκούς εθέρες, τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό και ένα σχετικό κανονισμό. Μέχρι στιγμής δυστυχώ δεν έχουμε σημειώσει επαρκή πρόοδο στο θέμα αυτό. Υπάρχουν κάποιες γεωγραφικές διαφορές. Είναι κατακαιρματισμένος ακόμη ο ευρωπαϊκός ουρανός δυστυχώ. Και στα θέματα των αερομεταφορών θα πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι. Ε, να αποφύγουμε τις καθυστερήσεις των πτήσεων, να μειώσουμε τις, εκπομπέ αερίων του θερμοκηπίου από τι αερομεταφορέ και να δούμε και το θέμα του ελέγχου τη ενέργεια κυκλοφορία. Σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των επιβατών των αερομεταφορών, ξέρω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει διαμορφώσει τη γνώμη του, που είναι πολύ σημαντική και θα τη λάβουμε υπόψη. Στόχο τη Φιλανδία είναι να καταλήξουμε σε μια γενική προσέγγιση στο Συμβούλιο, στο Συμβούλιο Μεταφορών του Δεκεμβρίου. Κάποιο αναφέρθηκε και στις διαπραγματεύσεις για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και το μηχανισμό συνδέοντα την Ευρώπη. Οι διαπραγματεύσεις για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο είναι βασική προτεραιότητα και μέλημά μας είναι να βρούμε μια ισορροπημένη λύση που θα λαμβάνει υπόψη τις νέες προτεραιότητες και μια ισορροπία μεταξύ των κλάδων ώστε να υλοποιήσουμε τους κοινού μας ευρωπαϊκούς στόχους. Η Φιλανδία έχει δεσμευθεί να προωθήσει την διεκπαιρέωση των συζητήσεων και του πλαισίου του ΠΙΔΕΛΤΑΠΗ μέχρι τα τέλη του έτου. Σε ό,τι αφορά την αυτοματοποίηση και την ψηφιοποίηση τη μεταφορέ, σίγουρα και τα δύο θέματα είναι σημαντικά για τη Φιλανδία, για τη Φιλανδική Προεδρία. Και το θέμα των ηλεκτρονικών εμπορευματικών μεταφορών είναι σημαντικό θέμα. Και τον Ιούνιο, όπως σας είπα, έχουμε καταλήξει σε γενική προσέγγιση στο Συμβούλιο και περιμένουμε την εντολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το ζητούμενο είναι να καταλήξουμε σε συνένεση μέχρι το φθινόπωρο, διευκολύνοντας την πρόοδο στα θέματα αυτά. Και να πω και λίγα λόγια για την αυτοματοποίηση. Πολλά είναι τα πλεονεκτήματά της. Ε, βελτιώνει την ε, ασφάλεια, μειώνει τις εκπομπές και ίσως ε, συμβάλλει στην καλύτερη διαχείριση του κυκλοφοριακού προβλήματος, της συμφόρηση. Βέβαια, κάτι τέτοιο προϋποθέτει έρευνα, ανάπτυξη προτύπων και φυσικά σημαντική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να καταλήξουμε στις σωστές αποφάσεις και να αποφύγουμε και τις επικαλύψεις. Θέσατε πολύ άριθμες ερωτήσεις. Πιστεύω ότι θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες να επανέλθουμε στα ζητήματα αυτά και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την Υπουργό Μεταφορών. Η Υπουργό Τουρισμού τώρα έχει να απαντήσει σε πολλές ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις. Να απαντήσω και εγώ λοιπόν στις ε, ερωτήσεις ε, για την ε, αηφορία στις ε, μεταφορές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό βεβαίως το θέμα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι η Προεδρία της Ρουμανίας ήταν πολύ σημαντική. Αναφέρθηκε και το θέμα της ε, ψηφιοποίησης, οπωσδήποτε Συμφωνία των Παρισίων και το πώς μπορούμε να επιτύχουμε τους ε, στόχους της. Με την ε, ψηφιοποίηση μπορούμε λοιπόν να προωθήσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη και να δώσουμε τις απαντήσεις στο θέμα της κλιματικής αλλαγής. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας θα προωθήσουμε λοιπόν το θέμα της ψηφιοποίησης και να αντιμετωπίσουμε και την κλιματική αλλαγή θα προσπαθήσουμε. Βεβαίως τα κράτη-μέλη μπορούν να προωθήσουν το θέμα και βεβαίως ε, είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε το πώς ε, ο τομέας των μεταφορών μπορεί να βοηθήσει στην ε, μείωση της κλιματικής αλλαγής. Θα ήθελα να τονίσω εδώ πως με την ψηφιοποίηση οι εταιρείες μεταφορών μεταβαίνουν προς την κυκλική οικονομία. Παραδείγματος χάρη υπάρχουν πολλές ευκαιρίες τις οποίες πρέπει να δούμε και ε, μπορούν να υπάρξουν και τοπικές ε, εξελίξεις. Μετά ε, κάποιος βουλευτής ρώτησε για τα ποδήλατα. Οπωσδήποτε είναι ένας τρόπος μεταφοράς βιώσιμος ε. αλλά αυτό είναι περισσότερο θέμα που είναι αρμοδιότητας ε, της Υπουργού Μεταφορών. Να αφαιρθώ σε αυτό το οποίο είπε ο κ. Κοντσούρ για την... Ε, για κουντουρά, με Για το θέμα της κοινωτικής στρατηγικής. Θα το δούμε οπωσδήποτε στο μέλλον με το χρονοδιάγραμμά μας μάλλον δεν θα απασχολήσει την Φιλανδική Προεδρία. Αλλά οπωσδήποτε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας θα προσπαθήσουμε να θέσουμε το ζήτημα αυτό. προτεραιότητά μας όπως σας είπα είναι η ψηφιοποίηση του τομέα των μεταφορών. Μετά, ε, κύριε Κοντουρά, πάλι κάτι για τον προπολογισμό. Έγιναν ε, κάποιες προτάσεις ε, ε, για έναν ξεχωριστό προπολογισμό στο πλαίσιο του ΠΔΠ. Ε, το Συμβούλιο θεωρεί ότι είναι σημαντικό ο τουρισμό, αλλά αντί ε, για να έχει έναν ξεχωριστό προπολογισμό είναι σημαντικό οι εταιρείε του τουρισμού να ωφεληθούν οριζόντια από τα διάφορα προγράμματα του ΠΔΠ με τον ίδιο τρόπο όπως οι άλλες εταιρείες σε άλλους κλάδους. Υπάρχουν διάφορα μέσα, το πρόγραμμα για την εσωτερική αγορά, τα γεωργικά ταμεία, το πρόγραμμα InvestEU για τις επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Euh, Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις, οι οποίες ε, νομίζω ότι θα οδηγήσουν και στο δεύτερο γύρο ερωτήσεων από τους βουλευτές για να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε. Και ξεκινάμε αμέσως από τον κύριο Ντελή. Να διευκρινίσω ότι δεν είναι εξάδελφός μου. Και γράφεται και με ένα L. Είμαστε στην αρχή της θητείας. Ε, κύριε Ντελή, εξηγώ σε όλους ότι δεν είμαστε εξαδέλφια. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ναι, δεν είμαστε συγγενείς, αλλά συνεργαζόμαστε καλύτερα γιατί δεν είμαστε συγγενείς ακριβώς. Γιατί ορισμένες φορές συγγενείς θυμώνουν ένας με τον άλλον. Ως, ε, όπως ανέφερε η αναπληρώτρια συντονιστής του ΕΛΚ, ε, εγώ θα μιλήσω για το πακέτο της κινητικότητας. Και Βλέπουμε ότι ασχολείστε με το θέμα της κινητικότητας. Δημιουργήθηκε όμως ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ των κεντρικών και περιφερειακών κρατών μελών. Και βάσει των όσων γνωρίζουν, ε, στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων του Συμβουλίου, η Φιλανδία διαδραμάτισε επικοδομητικό ρόλο και προσπάθησε να γεφυρώσει αυτό το χάσμα με κάποιο τρόπο, αλλά, ε, αλλά όλες οι προτάσεις οι οποίες ήταν πιο ισορροπημένες τελικά διαγράφησαν στο τέλος και τελικά τα μισά κράτη-μέλη έμειναν εκτός συμφωνίας. Και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τελικά ε, είχαμε μια αντίστοιχη κατάσταση. Οι συγητές από την προηγούμενη θητεία απλώς ε, αντέγραψαν λέξη προς λέξη το σχέδιο κειμένου της γενικής προσέγγισης και εμείς είμαστε νομοθέτες. Γι' αυτό ακριβώς ε, θεωρώ ότι στην προσπάθεια να καταλήξουμε σε μια ποιοτική νομοθεσία, η οποία θα οδηγήσει σε εύκολη εφαρμογή και ασφάλεια δικαίου για όλες τις πλευρές και όλους τους ενδιαφερομένους, θα πρέπει να επεξεργαστούμε λίγο καλύτερα αυτά τα θέματα, διότι είμαι πεπισμένος, ε, και δύο φράσεις ακόμα, ε, Είμαι πεπισμένο ότι τα κράτη-μέλη τα οποία έμειναν απ' έξω θα προσπαθήσουν ε, να βρουν ε, ε, λύσεις προσφεύγοντας ε, ακόμα και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πριν ακόμα την εφαρμογή τη νομοθεσία. Επομένω, αυτό θα οδηγήσει σε περαιτέρω προβλήματα στον τομέα. Και μόλι πριν από 10 λεπτά μα είπατε ότι προσπαθείτε να λάβετε υπόψη όλε τι απόψει και πραγματικά είμαι περίεργο πώς θα το καταφέρετε αυτό στην πράξη. Αλλά φυσικά εμείς είμαστε ανοιχτοί σε πιο ισορροπημένη προσέγγιση εδώ στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε κύριε Τελή, για αυτό το δεύτερο γύρο. Να υπενθυμίσω ότι ο καθένας από εσά έχει 1,5 λεπτό, διότι έχουμε 21 άτομα που έχουν ζητήσει το λόγο. Προς το παρόν δεν θέλω να περάσω το πρωί μου μαζί σας, το συγγνώμη και νομίζω ότι και οι υπουργοί έχουν και άλλα πράγματα να κάνουν. Συνεχίζουμε. Ο κύριος Μπεράντο, έχετε το λόγο. Για 1,5 λεπτό. Μάλλον πρέπει να συνηθίσω και με τους διάφορους τρόπους που προφέρει ο καθένας το ο επίθετό μου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τις υπουργού που είναι εδώ σήμερα, όχι μόνο σήμερα για τη συζήτηση, αλλά χθε ήσασταν και σε άλλες επιτροπές. Εγώ είμαι από μια περιοχή των κάτω χωρών που ε, ανήκει σε τρει ε, διευρωπαϊκούς διαδρόμους. Θα ήθελα να ξέρω πώ μπορούμε να επιταχύνουμε την υλοποίηση αυτών των ε, μεταφορικών δικτύων και να άρουμε το διοικητικό άχθο. Στο πρόγραμμα τη Προεδρία σα βλέπω ότι έχετε τονίσει ότι έχετε πρόθεση να εργαστείτε πάνω σε αυτά τα διευρωπαϊκά δίκτυα και παρά το γεγονό ότι το Κοινοβούλιο έχει ήδη εγκρίνει την πρώτη ανάγνωση για το ε, έξυπνο δίκτυο μεταφορών, το Συμβούλιο ακόμα δεν έχει καταλήξει κάποια θέση. Έχω δύο ερωτήσεις λοιπόν. Πρώτον, τι προτεραιότητα έχει ε, το θέμα αυτό στην Προεδρία σας και δεύτερον, τι χρονοδιάγραμμα περιμένετε να έχουμε στο Συμβούλιο, πότε μπορούμε να περιμένουμε μια θέση του Συμβουλίου ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε και τις διοργανικές διαπραγματεύσεις στη συνέχεια. Καλή τύχη για την Προεδρία σας και φυσικά προσβλέπω και στη συνεργασία μας το επόμενο εξάμεινο. Ευχαριστώ. η κυρία Λισαντό. Για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, Υπουργοί, ο τομέας των μεταφορών, είναι, ο τουρισμού συγγνώμη, είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη χώρα μου. Είναι η χώρα με του περισσότερου επισκέπτε, ε, πάνω από 80 εκατομμύρια επισκέπτε πέρσι και εγώ είμαι από μια τουριστική περιοχή τη Γαλλία. Θα ήθελα λοιπόν να σα ρωτήσω κάτι για ένα τομέα που είναι σε πλήρη ανάπτυξη, τον τουρισμό κρουαζιέρας, ε, που αφορά και αρμοδιότητα ε, και των δύο θεμάτων, και τις μεταφορέ και του τουρισμού αυτέ τι επιτροπέ. Αυξήθηκε κατά πολύ ο τουρισμό κρουαζιέρα και η χώρα χώρα που έχει 32 μεγάλους προορισμούς ε, και έχουμε πάνω από 90 λιμάνια στον κόσμο, θα θέλαμε ε, να μας πείτε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης όπως και όλες οι παράκτιες ε, χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας ενδιαφέρουν οι επενδύσεις και ο σεβασμός προς το περιβάλλον. Θα πρέπει λοιπόν να χρηματοδοτήσουμε μια στρατηγική ανάπτυξη του τουρισμού κρουαζιέρας με τη βελτίωση της υποδοχής ε, στους θερματικούς σταθμούς ε, και στις πόλεις λιμάνια, αλλά να βρούμε και έναν τρόπο να χρηματοδοτήσουμε την κατασκευή ιδίων σκαφών. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη επίσης ε, την ε, ηλεκτροδότηση των σκαφών, ε, την απόρριψη των απορριμμάτων και για να έχουμε ένα κατάλληλο καθαρό τουρισμό σίγουρα θα έχουμε δυσκολίες. Πώς μπορείτε να βοηθήσετε λοιπόν αυτό τον ουσιαστικό τομέα με τους πόρους που χρειάζεται. Ευχαριστώ και σας ευχαριστώ που σέβεστε το χρόνο. Ο κύριος Δενίλσεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω σου ειδικά. Κύριε Υπουργέ, Υπουργή, μία ερώτηση η οποία αναφέρθηκε ήδη εδώ για το θέμα της κινητικότητας, το καμποτάζ και ούτω καθεξής. και το θέμα των αποσπάσεων. Η οδηγία αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική για μας. Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα μεταφορών το οποίο θα είναι κοινωνικά βιώσιμο, ε, θα πρέπει να υπάρχουν συνθήκες εργασίες οι οποίες θα πρέπει ε, να εγγράφονται σε αυτή την οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων. Θα ήθελα να ξέρω κατά πόσον η Προεδρία σας λοιπόν σκοπεύει να ξεκινήσει τριμερή διάλογο για το θέμα αυτό στο πακέτο της κινητικότητας διότι υπάρχει και μία ακόμα έννοια. Θα πρέπει να εφαρμόσουμε και όλα αυτά που έχουν εγκριθεί. Σκοπεύετε να τα εφαρμόσετε όλα αυτά τα οποία έχουν μέχρι τώρα εγκριθεί. Στο πρόγραμμα εργασία αναφέρεστε επίση τι αρχέ εργασία. Θέλετε ή όχι να συνεχίσετε προ αυτή την κατεύθυνση. Ε, και να μας πείτε και τι δυνατότητες υπάρχουν σε θέματα οδικών μεταφορών ε, με τις παρούσες αρμοδιότητες θα μπορέσετε να βρείτε κάτι για τις ε, οδικές μεταφορές ή όχι. Ε, πιστεύετε ότι η ψηφιοποίηση των οδικών μεταφορών είναι δυνατές. Ευχαριστώ. Η κυρία Τεπαρβό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητές Υπουργοί, Σάννα Μαρίν και Κατρίν Κουλμούνη. Σας ευχόμαι καλή επιτυχία για να προωθήσετε ακριβώς αυτή την μετάβαση στον τομέα των ε, μεταφορών. Έχω μία ερώτηση που αφορά τα δικαιώματα των επιβατών σιδηροδρόμων. Ακόμα δεν έχει περάσει το πακέτο από το Συμβούλιο. Το Κοινοβούλιο έχει ψηφίσει μία ξεκάθαρη θέση και ζητάει βελτίωση αυτών των δικαιωμάτων για να αναγνωριστεί ακριβώς ε, αυτός ο τρόπος μετακίνησης που είναι πολύ φιλικός προς το κλίμα και να γίνει πιο ελκυστικός. Στο Συμβούλιο όμως δεν συμβαίνει κάτι άλλο. Τι σκοπεύετε να κάνετε ως Προεδρία στο μέλλον έτσι ώστε να ανταποκριθεί στο όνομά του αυτός ο κανονισμός και να υπάρχουν και νέοι τύποι εισιτηρίων με ανοιχτά δεδομένα και βεβαίως να έχουμε και καλύτερη πρόσβαση ατόμων με κινητικές ε, δυσκολίες. Κάτι στο οποίο η Φιλανδία έχει κάνει αρκετά καλά βήματα. Σας ευχαριστώ. Κύριε Σολιβιέ. Έχετε 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ Μεταφορών, άκουσα την ε, τεχνική και μελλοντοστραφή σας παρέμβαση, αλλά μου φάνηκε λίγο κρύα, για να μην πω παγωμένη. Μας μιλήσατε για δεδομένα, για ψηφιοποίηση, για αυτοματοποίηση, για απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα. Μέσα σε 10 λεπτά βέβαια αναγνωρίζω ότι δεν μπορεί να καλύψει κανείς τα πάντα. Αλλά υπάρχει ένα θέμα που το αμελήσατε και κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σημαντικό. Το ανθρώπινο στοιχείο, ο ανθρώπινο παράγοντας πίσω από τις αποφάσεις, τις εκθέσεις, τις οδηγίες υπάρχουν άνθρωποι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι έβαλε ως ακρογωνία της εποχής της ε, πολιτικής μεταφορών την απόσπαση εργαζομένων. Οπότε διαρωτόμαστε αν ε, έχει τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Μιλήσατε κάπω ασαφώ για τα κοινωνικά συμφέροντα. Τι γίνεται όμω με τα κοινωνικά συμφέροντα των αποσπασμένων εργαζομένων. Και υπάρχει μάλλον το ζήτημα τη αξιοπρέπεια. Στη Γαλλία βλέπουμε Πολωνούς ή Ρουμάνους ε, φορτηγατζίδες που μένουν ουσιαστικά, που ζουν στους χώρους στάθμευσης, ε, που κοιμούνται στις, ε, στους θαλάμους των φορτηγών. Είναι πραγματικά ε, φυλακισμένοι των, οδικών μεταφορών, φυλακισμένοι στα συνταλίκες τους. Πώ θα λάβετε υπόψη λοιπόν τον κοινωνικό αντίκτυπο των δικαιωμάτων των ε, αποσπασμένων εργαζομένων στη διάρκεια της πολιτικής που θα ακολουθήσετε ως Φιλανδική Προεδρία. Ευχαριστώ. Χωρί μικρόφωνο δυστυχώ. η πρόεδρο. Η κυρία Βιρκούναν. Σα ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ ε, τη συνάδελφα που μου έδωσε τη θέση της, ε, γιατί πρέπει να φύγω για το αεροδρόμιο και θα ήθελα και εγώ ως η μοναδική Φιλανδέζα της Επιτροπής να μην χάσω την ευκαιρία να καλωσορίσω τις δύο Φιλανδές υπουργού. Ευχαριστώ τις δύο υπουργού που μας παρουσίασαν τις προτεραιότητες της Φιλανδικής Προεδρίας και μια και οι συνάδελφοι έθεσαν πολύ σημαντικέ ερωτήσει για την κλιματική πολιτική που είναι από τι σημαντικότερε προτεραιότητε τη φιλανδική προεδρία και το ε, πακέτο κινητικότητα ήδη με κάλυψαν. Το πακέτο κινητικότητα ίσω είναι η πιο περίπλοκη νομοθετική πρόταση που έχουμε επιτάπητο και ζητούμενο είναι ισορροπημένε λύσει και στο πακέτο αυτό. Εγώ έχω μία ακόμη ερώτηση για την Φιλανδική Προεδρία. Μία από τις κρίσιμες αποφάσεις που θα κληθούμε να λάβουμε θα είναι η απόφαση για τις δημοσιονομικές προοπτικές, το μελλοντικό πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο και τέθηκαν αρκετές ερωτήσεις για το θέμα αυτό και ιδιαίτερα για το μηχανισμό συνδέοντας την Ευρώπη. Πολύ σημαντικό θέμα για την Επιτροπή μας και θα έχει κέρια σημασία για την ανάπτυξη ε, σύγχρονων και ε, ευφυών ε, υποδομών μεταφορών για να έχουμε πραγματικά έξυπνες και αποδοτικέ συνδέσει. Ήδη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στι αρχέ του έτου κατέληξε στην απόφαση να ενισχύσει το τμήμα κινητικότητα του μηχανισμού συνδέοντα την Ευρώπη. Η Φιλανδική Προεδρία είναι υπέρ τη ενίσχυση του τμήματο κινητικότητα του μηχανισμού συνδέοντα την Ευρώπη στι διαπραγματεύσει για το πει. Και πώς πιστεύετε ότι το, ο μηχανισμός αυτός θα βελτιώσει πραγματικά τις διασυνδέσεις στην Ευρώπη και πώς θα προσελκύσει επενδύσεις για να έχουμε πραγματικά ευφυείς υποδομές στις μεταφορές της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ. Εσείς λίγο αργότερα. Γιατί πρέπει να σεβαστούμε τις ισορροπίε μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Να μην έχουμε ερωτήσεις ε, μόνο από μία πολιτική ομάδα. Η κυρία Γκουτεζάρ, πού είστε παρακαλώ. 1,5 λεπτό κι εσείς. Σας ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να καλωσορίσω τις δύο υπουργούς στην ε, Επιτροπή Μεταφορών. Το πρόγραμμα ε, της ε, Φιλανδικής Προεδρίας ε, μας δίνει σημαντικές κατευθυντήριες γραμμές για πολλές ε, πολιτικές και για την πολιτική των μεταφορών. Στο έγγραφο εργασίας που υπέβαλε στο Συμβούλιο η Φιλανδική Προεδρία αναφέρεται και σε κάποια ζητήματα της ναυτιλίας. Αναφέρεται για παράδειγμα στη συνεργασία με το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό προκειμένου να προωθηθεί ο ρόλος της Ευρώπης παγκοσμίω και να έχουμε βιώσιμες και αυτοματοποιημένες και ναυτιλιακές μεταφορές. Αυτό που με ενδιαφέρει συγκεκριμένα είναι τι ε, ρόλο θα δώσετε στην πολιτική για την ναυτιλία στο πλαίσιο της γενικής στρατηγικής ε, για τις μεταφορές. Επίσης, ε, τι δράση θα αναλάβετε για να προωθήσετε μια αποτελεσματική ναυτιλιακή πολιτική με περισσότερη διασυνδεσιμότητα, με αποτελεσματική και ευφύ διασύνδεση μεταξύ των νησιών και των παράκτειων περιοχών. Γιατί και εγώ από νησί κατάγομαι και γνωρίζω πόσο σημαντικές είναι οι συνδέσεις μεταξύ των νησιών. Ποια είναι λοιπόν τα σχέδια της Φιλανδικής Προεδρίας για την βελτίωση της διασυνδεσιμότητας στην αυτιλία. Σας ευχαριστώ. Κύριε Ροντρίγκες. Έχετε κι εσείς 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ πρώτα απ' όλα να καλωσορίσω τις δύο υπουργούς της Φιλανδικής Προεδρίας και να ευχηθώ καλή επιτυχία. Είμαι βεβαία ότι θα έχουμε αγαστή συνεργασία, γιατί η επιτυχία της Φιλανδικής Προεδρίας θα είναι κοινή επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω τρεις ερωτήσεις. Σε ό,τι αφορά τις μεταφορές, μας είπατε πόσο Σημαντικό είναι να ενισχύσουμε τα δικαιώματα των καταναλωτών. Συμφωνούμε και εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το θέμα αυτό. Σε ό,τι αφορά τώρα τους ε, χρήστες, τους επιβάτες ε, low cost ε, αεροπορικών εταιριών, πολύ συχνά χρησιμοποιείται η ψηφιοποίηση ως φραγμός για να αποτρέψουν τους επιβάτες να ασκήσουν τα δικαιώματά τους και να κάνουν τις διεκδικήσεις τους πώς μπορείτε συγκεκριμένα να ενισχύσετε τα δικαιώματα των επιβατών, ε, κυρίως τέτοιων ε, ε, αεροπορικών εταιριών χαμηλού κόστους. Σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, χάρη στην ψηφιοποίηση έχουμε όλο και μεγαλύτερη χρήση των διαμερισμάτων και των κατοίκων στον τουρισμό. Και μερικές φορές υπάρχουν προβλήματα σε διάφορες χώρες με τους χρήστες και τις πολιτικές του τουρισμού. Πρόκειται να προτείνεται μια μεγαλύτερη ομογενοποίηση της κατάστασης, να γίνει πιο ομοιόμορφη στα κράτη-μέλη και πότε. Σε ό,τι αφορά τις κλιματικές αλλαγές ε, και την αυτιλία, πώς θα καταφέρουμε να διαφυλάξουμε τους ωκεανούς μας, τι προτάσεις ε, θα κάνετε για την αυτιλία ώστε να σταματήσει αυτή η ρήπανση των ωκεανών. Σας ευχαριστούμε κυρία Ροτρίγκες. Κυρία Ουκασεύσκα, ήρθε και η δική σας σειρά. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω τις δύο υπουργού και ελπίζω η Φιλανδική Προεδρία και οι γυναίκες εκπρόσωποι της να προωθήσουν πολύ πιο αποτελεσματικά αυτό το πακέτο κινητικότητας. Ε, λαμβάνοντας υπόψη και τα οικονομικά σκέλη, αλλά και τις αξίες και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η ελεύθερη διακίνηση προσώπων και εμπορευμάτων σε μια ενιαία εσωτερική αγορά. Έχω μια ερώτηση λοιπόν. Πώς σκοπεύει η Φιλανδική Προεδρία να συνδυάσει τις ε, αξίες και τις αρχές της ενιαίας αγοράς με τον περιορισμό των δραστηριοτήτων ε, στα πλαίσια της άσκησης των υπηρεσιών των ενδομεταφορών του ΚΑΠΟΤΑΣ ή στην περίπτωση της απόσπασης των εργαζομένων. Πώς θα συνδυάσουμε τον περιορισμό του ΚΑΠΟΤΑΣ με τις βασικές ε, αρχές μας και τις προσπάθειες να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Γιατί ακούσαμε από χώρες της ε, Ανατολικής Ευρώπης ότι ουσιαστικά δημιουργούνται προβλήματα ανταγωνιστικότητας και αυτό γίνεται, υποτίθεται ε, για να διορθωθούν κάποιες ανισότητες, αλλά δεν θα πρέπει να έχουμε στρέβλωση ανταγωνισμού. Επίσης, με το Brexit τι θα γίνει, πώς θα επηρεάσει το Brexit ε, τις υπηρεσίες των μεταφορών. Ε, και τα θέματα της ε, ναυτιλίας. Έχουμε τεράστιες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα από τις ναυτιλιακές μεταφορές. Αυτό δεν το λέει κανείς. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πίτερ Λούγκριν έχει το λόγο. Για 1,5 λεπτό κι εσείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω κάποια ερώτηση. Θα ήθελα απλά να σας υπενθυμίσω ότι το πακέτο κινητικότητας έχει πολύ μεγάλη σημασία. Υπάρχουν πολλά προβλήματα σε διάφορους δρόμους στην Ευρώπη. Το πακέτο δεν έχει ολοκληρωθεί. Και βεβαίως αυτό δεν είναι μπομφή προς τον συνάδελφο τον Ισμαήλ που έχει κάνει εξαιρετική δουλειά αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, να έχουμε σαφείς κανόνες, να δημιουργηθούν οι συνθήκες ε, για να έχουμε μια σοβαρή λειτουργία και δεν είναι δυνατόν βεβαίως να τα αφήσουμε όλα αυτά μόνο στους συμμετέχοντες στην αγορά. Τέλος θα ήθελα να φέρω και το περιβάλλον γιατί οι συγκοινωνίες αποτελούν σημαντικό κομμάτι των εκπομπών στη Σουηδία και στη Φιλανδία υπάρχουν ε, μεγαλύτερα φορτηγά από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εντάξει, αυτό δεν είναι πρόβλημα βεβαίω. Αν δούμε πόσα φορτηγά μετακινούνται π.χ. από τη Βόρεια Γερμανία στη Νότια Γερμανία. Οπότε είναι διαστρεβλωμένο να λέμε ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε μεγαλύτερα φορτηγά. Εξάλλου είναι καλύτερα για το περιβάλλον. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Λιμπεράτσκι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υπουργοί, σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Πρώτα απ' όλα, πακέτο κινητικότητας. Αυτός είναι ένας καλός λόγος που μπορεί να διχάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι θα κάνετε για να υπάρξει ξανά συνοχή. Κατόπιν ε, τα περιφερειακά πακέτα, ειδικά ο διάδρομος ε, προς την Βαλτική. Μπορείτε να μας βοηθήσετε να γίνει βιώσιμο αυτό το έργο με έναν καλό συντονιστή. Αναμένουμε να δοθεί το πράσινο φω για του σιδηροδρόμου. Πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο κατόπιν. Ε, μου αρέσει η ιδέα που έχετε για εξυγχρονισμό, πιο αποτελεσματικέ υποδομέ, αλλά γνωρίζουμε ότι πάντα υπάρχει έλλειψη χρημάτων. Αναμένετε τέτοιε δυνατότητε όπω π.χ. την χρήση του σχεδίου το Juncker και τη σχετική χρηματοδότηση μέσω ομολόγων έργων ε, ή συμπράξεων δημοσίου ιδιωτικού τομέα του μέσου συνδέοντα στην Ευρώπη να συνδυαστούν όλες οι πιθανές πηγές καρματοδότησης έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή στις ευρωπαϊκές πόδες Και 10 ε, νωρίτερα τελείωσα κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Λιμπεράτσκι. Ο κύριος Λούτκεν. Συγχαρητήρια και θερμό καλωσόρισμα στις δύο υπουργούς. Σίγουρα θα νιώθετε πολλές στιγμές χαράς αλλά και απογοήτευσης. Ε, και εγώ διατέλεσα υπουργό μεταφορών και συμμετείχα δύο φορέ σε τέτοια συμβούλια μεταφορών. Και τα έχω βιώσει και εγώ αυτά. Μιλήσατε για βιωσιμότητα, για κλίμα, πολύ σημαντικέ προκλήσει όλε αυτέ. Αλλά ελάχιστα μιλήσαμε για απασχόληση, ελάχιστα μιλήσαμε για την οικονομία και πολύ ακροθυγό και για τα κοινωνικά ζητήματα ενώ και ο τομέας μεταφοράς και ο τομέας ε, τουρισμού είναι τομείς που εξασφαλίζουν βιοπορισμό πολλών εκατομμυρίων πολιτών και επιχειρήσεων. Επίσης, έχουμε κάποιες ζώνες που είναι εγκλωβισμένες στην Ευρώπη. Δεν έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ, στις νέες τεχνολογίες. Πολύ ωραία να μιλάμε για ψηφιοποίηση, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν ε, υποδομές ε, ε, για να μπορούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στους παρόχους, αλλά μερικές φορές υπάρχει και ένας τέτοιος εγκλωβισμός και απομόνωση από τις δημόσιες μεταφορές και για τις επιχειρήσεις και για τους πολίτες. Οπότε υπάρχει κατεπίγουσα πολιτική και οικονομική ανάγκη να εξασφαλίσουμε τέτοια προσβασιμότητα. Ε, και μερικές φορές δυστυχώς ε, επικρατούν κάποιες εξτρεμιστικές απόψεις. Ποια είναι ε, τα σχέδιά σας για να εξασφαλίσουμε πρόσβαση σε εκατομμύρια πολίτες που έχουν αποκλειστεί μερικές φορές από το, τις μεταφορές και την οικονομία. Ναι, σας υπενθυμίζω όμως ότι η μάχη για το κλίμα είναι μάχη και υπέρ της απασχόλησης. Και είναι σημαντικό να το διευκρινίζουμε αυτό στην Επιτροπή μας. Ο κύριος Σκοτ. Ένα, ενάμιση λεπτό. Okay, uh, thank you. Ευχαριστώ. Σας καλωσορίζω Καλωσορίζω την Προεδρία σας και όπως ε, οι άλλοι νεαροί, Σκανδιναβοί, η Γκρέτα Τόνμπρι τι θα, τι θα κάνετε κι εσείς για να βοηθήσετε στην σαφήνεια του μηνύματος για να επιτύχουμε ουδετερότητα ως προς τον άνθρακα μέχρι το 2050. Χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους του Λονδίνου για να σταματήσουν την κίνηση, για να πούνε ότι πρέπει αυτό να γίνει μέχρι το 2025. Η Βρετανική κυβέρνηση τώρα βέβαια στοχεύει στο 2050, αλλά υπάρχουν κόμματα που πιέζουν για το 2030. Ακούγονται λοιπόν όλοι αυτοί οι αριθμοί. Τι θα κάνετε για να ξεκαθαρίσει το θέμα με τις αντιφατικές πληροφορίες που ακούγονται και δυστυχώς δεν σημειώνεται πρόοδο στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Έχουν γίνει λίγα πράγματα για να επιτύχουμε την ουδετερότητα ως προς το κλίμα. Λοιπόν, τι θα κάνετε για να είναι σαφέστερο το μήνυμα προς τους Ευρωπαίους εκείνους που αισθάνονται αποξενωμένοι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά και κάτι άλλο. Μπορείτε να μας δώσετε κάποια ξεκάθαρα βήματα στρατηγικά να μας πείτε ποια είναι τα βασικά εμπόδια για να επιτύχουμε κάτι τέτοιο και σας παρακαλώ να είστε ειλικρινείς. Σας ευχαριστώ. Για... Σας ευχαριστούμε για το σαφέστατο σας μήνυμα. Συνεχίζουμε. Ο κύριος Νάβακα, πού είστε, καλημέρα σας. Έχετε το λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι λακωνικός. Να σας καλωσορίσω αγαπητές ε, Υπουργοί. δεν μπόρεσα να αντισταθώ στην εσωτερική μου επιθυμία να μιλήσω για το πακέτο της κινητικότητας, παρόλο που μου υποσχέθηκα ότι δεν θα το κάνω. Εσείς ε, ε γνωρίζετε ότι μας έχει διχάσει ε, σε σημείο που η Επιτροπή δεν μπόρεσε να έχει διαθέσει για το θέμα αυτό. Μας δίχασε λοιπόν πάρα πολύ πέραν το γεγονότος ότι δηλώσατε ότι ελπίζετε να το προχωρήσετε, πώς ε, σκοπεύετε ε, να πείσετε τους πάντες να συμμετέχουν για το θέμα αυτό, διότι όπως γνωρίζετε όλοι έχουμε το ίδιο πάθος για τις μεταφορές ε, και θα ήταν κρίμα αν δεν εκπροσωπούνται οι μισές χώρες στο θέμα αυτό. Πώς πιστεύετε λοιπόν ότι θα γίνει αυτό, πώς θα μπορέσουμε να πείσουμε τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής να ασχοληθούν με το θέμα αυτό και να συμμετέχουν. Επίσης, ε, οι συνδυασμένε μεταφορές, διότι η πρώτη μου ευθύνη εδώ στην Επιτροπή είναι να είμαι σκιώδης ε, ε, εισηγητή για τις συνδυασμένε μεταφορές. Τι φιλοδοξίες έχετε εσεί λοιπόν για το θέμα αυτό, πώς βλέπετε να προχωρά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. 15 δευτερόλεπτα οικονομία σας έκανα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βιτάνοφ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμοι Υπουργοί, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα και εγώ να απευθύνω την ερώτησή μου προς την Υπουργό Μεταφορών, αλλά θα συνεχίσω στα βουλγαρικά, μου επιτρέπετε. Όσον αφορά τους φιλόδοξους στόχους που θέσατε, η προτεραιότητα της μείωσης των εκπομπών ε, και η ψηφιοποίηση είναι προτεραιότητες ε, με τις οποίες συμφωνούμε. Ελπίζουμε όμως ότι θα είστε ε, ειλικρινείς διαμεσολαβητής στη διαπραγμάτευση για τα θέματα αυτά, για το πακέτο για την κινητικότητα. Ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ λεπτό το θέμα αυτό για τις περιφερειακές χώρες. Στη Βουλγαρία δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να μας πετάξουν έξω από την εσωτερική εξωτερική αγορά. Ε, ανησυχώ ιδιαίτερα για το θέμα αυτό και το ενδεχόμενο μεγάλο τμήμα των προσανατολισμών ε, του διεθνούς, ε, των διεθνών μεταφορών να βρεθούν να χάνουν δουλειέ στη Βουλγαρία γιατί δεν μπορούν να συμμετέχουν. Πολλέ από τι επιχειρήσει στην Βουλγαρία είναι μικρομεσαίε επιχειρήσει, οικογενειακέ επιχειρήσει, επομένω η μόνη πηγή εισοδήματο για μια ολόκληρη οικογένεια ορισμένε φορέ. Ε, τι σκοπεύετε να κάνετε λοιπόν για να μην χρεοκοπήσουν και να μην χάσουν τη δουλειά τους αυτοί οι άνθρωποι. Και επίσης, ε, στην προηγούμενη θητεία του Κοινοβουλίου υπήρχαν κάποιες αποφάσεις οι οποίες αντιβαίνουν με το στόχο της Προεδρίας όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών η επιστροφή κενών οχημάτων στις χώρες ε, καταγωγής ή ε, στις χώρες που είναι γεγραμμένα τα οχήματα. Πώς βλέπετε λοιπόν αυτή την αντίφαση ε, με το χάσμα Ανατολής δύση και την πράσινη οικονομία και επίση τι άποψη έχετε εσείς για να προχωρήσετε το πακέτο κινητικότητας. Θεωρείτε ότι το κείμενο που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ισορροπημένη βάση για το μέλλον. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φρίγκο. ste Σας καλωσορίζω, παρουσιάσατε τις προτεραιότητες σας. Αυτό το οποίο με χαροποιεί είναι ότι ε, πρώτες ε, προτεραιότητες είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Ε, πάρα πολύ θετικό αυτό και τα ίδια μας είπε και η κυρία Ούρσουλα Φαντελάιν Βεβαίω, ε, αυτά δεν γίνονται σε έξι μήνες της ε, Προεδρίας ε, αλλά γνωρίζουμε ότι μετά ακολουθεί η Κροατία και έχετε αυτή την τρίπλη Προεδρία, Ρουμανία, Φιλανδία, Κροατία και εκεί πέρα μπορεί να γίνει κάτι οπότε είστε σε επικοινωνία με την Κροατία έτσι ώστε η προστασία του περιβάλλοντος να γίνει μια βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαι από την Κροατία, γι' αυτό τα ρωτάω αυτά. Η κυρία Γκραπίνη, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας ε, στην Προεδρία και να καλωσορίσω και τη Φιλανδική Προεδρία και να τους ευχηθώ ότι καλύτερο. Θα ήθελα να απευθύνω μια ερώτηση για τη διασύνδεση των σιδηροδρόμων. Τι προθέσεις έχετε προκειμένου να βελτιώσουμε τη διασύνδεση των σιδηροδρόμων, δεδομένου ότι στις περιφερειακές χώρες οι σιδηρόδρομοι ε, είναι σε ικτρή κατάσταση και δεν υπάρχει σύνδεση με περιοχές ε, των δυτικών χωρών. Έχετε λοιπόν και την καυτή πατάτα το πακέτο κινητικότητας και ανάλογα με τον τρόπο που θα εξελιχθεί θα μπορέσουμε ίσως να παρέχουμε ισότιμους αέρους ανταγωνισμού στον τομέα αυτό. Εγώ είμαι μέλος και της Επιτροπής ΣΥΜΚΟ. Πρέπει λοιπόν να σεβαστούμε και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Ξέρετε όμως ότι υπάρχει η σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα κράτη-μέλη να υπάρχουν ασφαλείς χώροι και στέγαση για τους εργαζομένους. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Επιπλέον, το πακέτο για την κινητικότητα προβλέπει υποχρέωση των οδηγών ε, να ε, υποχρέωση συγγνώμη, να προσφέρεται στέγαση στους οδηγούς. Και υπάρχουν φυσικά και θέματα ασφάλειας, ε, ληστείες, ε, κλοπή εμπορευμάτων κλπ. Πώς μπορείτε λοιπόν να ολοκληρώσετε αυτό το αμφιλεγόμενο πακέτο για την κινητικότητα, το οποίο έχει ψηφιστεί ε, με παραβίαση των κανόνων. Ξέρετε ότι η κατάσταση ήταν πολύ πολύπλοκη. Έγινε μία ψήφος, ε, ψηφοφορία μπλοκ παρά το γεγονός ότι αυτό δεν συνάδει με τον κανονισμό του Κοινοβουλίου. Υπάρχει λοιπόν ένα φορολεγόμενο πακέτο και εσείς είστε αρμόδιοι γι' αυτό. Ξέρουμε ότι η Φιλανδία υπερψήφισε το πακέτο στο Συμβούλιο, αλλά δεν καταφέρατε να εκπληρώσετε και τις ελπίδες ε, για τη μείωση των εκπομπών. Ε, αν ε, επιστρέφουν κενά τα οχήματα χωρίς εμπορεύματα, πώς θα προχωρήσει αυτό. Ο κύριος Μιλάζο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και τις υπουργούς σου για τη σημερινή τους παρουσία. Εγώ είμαι από τη Σικελία, περιοχή που ε, ε, ε, λαμβάνεται στο διάδρομο της Μεσογείου και μεταξύ των προτεραιοτήτων για τις επενδύσεις λείπει οποιαδήποτε αναφορά στις νησιωτικές περιοχές και μάλιστα στη Σικελία πιο συγκεκριμένα. Ε, στο Συμβούλιο, στις διαπραγματεύσεις, ε, ε, λέγεται ότι θα πρέπει να συζητηθεί το ποσό για κάθε κεφάλαιο για να δούνε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια αυτά για την ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών δικτύων. Στην περιοχή μου λοιπόν, την οποία εκπροσωπώ, η Φιλανδική Προεδρία σκοπεύει να προχωρήσει στη διαπραγμάτευση και να δώσει όθηση για την έγκριση του κανονισμού που θεσπίζει τον κανονισμό για να διασυνδεθεί η Ευρώπη. Διότι ο, ο, ο διάδρομος αυτός λέγεται ε, διάδρομος Σκανδιναβίας Μεσογείου. Διότι θα υπάρχει συνδεσιμότητα μόνο αν μπορέσουμε να συνδέσουμε τη Βόρεια Ευρώπη με ανθρώπους που βλέπουν στη Μεσόγειο και αυτό μπορεί να γίνει μόνο εάν το συνδέσουμε με την Νότια Ευρώπη. Δεν χρειάζεται να σας πω τι αντίκτυπο θα έχει στην υποστήριξη ε, και στο εμπόριο και στις θέσεις εργασίας, ακόμα και στον τουρισμό, αλλά κυρίως και για το περιβάλλον. Περιμένουμε λοιπόν από την Προεδρία σας μια σαφή δέσμευση, αποφασιστική και συγκεκριμένη για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λύρη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι αντιπρόεδρος ε, της Επιτροπής αυτής ε, που είναι αρμόδια για τον τουρισμό και ήμουνα και στην προηγούμενη θητεία. Αντιλαμβάνομαι πόσο δύσκολο είναι να ασχολείστε με τόσα πολλά ζητήματα. Ήμουν και υφυπουργό. Το καταλαβαίνω λοιπόν. Ταυτόχρονα όμω έχω την αίσθηση ότι κάτι λείπει η ακρόαση αυτή στην επιτροπή αυτή. Μου φαίνεται ε, ότι έχει παραμελήσει τελείως τον ε, τουρισμό. Και όμως έχουμε σε αυτή την επιτροπή τρεις-τέσσερις πρώην υπουργού ε, τουρισμού που ε, βρίσκονται εδώ ακριβώς γιατί θέλουν να προωθήσουν τον ε, τουρισμό στην Ευρώπη. Δεν έχουμε τόσο πολλές νομοθετικές αρμοδιότητες στον τομέα του τουρισμού. Αλλά εάν δεν προσέξουμε και δεν προωθήσουμε τον τουρισμό θα έχουμε πολλά προβλήματα. Γιατί χωρίς τουρισμό και χωρίς μέτρα που θα προωθούν τον τουρισμό ή όλη αυτή η αρχιτεκτονική του τουρισμού θα καταρρεύσει. Υπάρχουν πολλά προβλήματα αλλά και ευκαιρίες βεβαίως. Ε, έχω απευθύνει μια επιστολή προς την Προεδρία. Σας παρακαλώ να την δείτε. Ζητάμε αλλαγές στο ΠΔΠ και έναν ξεχωριστό προϋπολογισμό για τον ε, τουρισμό. Σας ευχαριστώ. Κυρία Μέτς, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και τις δύο υπουργούς ε, για το χρόνο που μας αφιέρωσαν. Δύο ερωτήσεις έχω. Πώς σκοπεύετε να βελτιώσετε τις διασυνδέσεις μεταξύ των διαφόρων πόλων της Ευρώπης γιατί αν συγκρίνουμε με άλλες χώρες, για να πάει κανείς από το Τόκιο στην Οζάκα, ε, στην Ιαπωνία, το καταφέρει μέσα σε δύο ώρες, δεν χρειάζεται να αλλάξει τρένο. Ενώ εγώ για να πάω από το Λουξεμβούργο στο Βερολίνο, που είναι ίδια περίπου απόσταση, χρειάζομαι εννέα ώρες και τρεις ανταποκρίσεις. Πρέπει να αλλάξω τρεις φορές τρένο. Τι σκοπεύετε να κάνετε λοιπόν για να βελτιώσετε τις ε, διασυνδέσεις και να προωθήσετε και τα τρένα υψηλής ταχύτητας για να βελτιώσουμε ε, το χρόνο γιατί όπω σα είπα από το Λουξεμβούργο να έρχομαι στι Βρυξέλλε θέλω τρει ώρε. Μ' αρέσει να βλέπω τα μικρά χωριά και το ειδηλιακό τοπίο, αλλά προτιμώ να έρχομαι πιο γρήγορα. Θέλουμε τρένα υψηλή ταχύτητα. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν να επανέλθουμε και στα νυχτερινά τρένα που είχαμε στο παρελθόν, που είναι και πολύ ευχάριστο να ταξιδεύει κανεί μπορούμε να αναλάβουμε κάποιες δράσεις για να προωθήσουμε και πάλι την ανάπτυξη των νυχτερινών τρένων, γιατί τα νυχτερινά δρομολόγια έχουν εκλείψει σχεδόν. Επίσης, πώς σκοπεύετε να συνδέσετε τις μεταφορές και τον τουρισμό, ώστε σε όλα τα τερματικά, όλοι οι σταθμοί παντού να είναι προσβάσιμοι σε όλα τα άτομα, ακόμη και με αναπηρίες, για να μην χρειάζεται να ζητά κανείς ειδικό κλείδι για να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα σε έναν σταθμό. Γιατί αν όλοι είχαν υπογράψει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα άτομα με αναπηρίες, κάτι που δεν έχει γίνει δυστυχώς, θα είχαμε ε, σε όλες τους σταθμούς και τους σιδηροδρομικούς και στα άλλα τα τερματικά δυνατότητα χρησιμοποίηση και πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες. Και ενώ και τους τυφλούς, τους κοφούς και άλλες αναπηρίες. Ε, λεπτό, η ε, κυρία Βιλτερά. Ε, μπαραντίκα, συγγνώμη. Ε, λυπάμαι που έλειψα κάποια στιγμή γιατί παρουσιάσαμε στον τύπο ένα πρόγραμμα για τον τουρισμό που συνδέεται με το έρασμος ε, ΣΥΝ, το ενισχυμένο έρασμος. Επίσης, μιλούμε για έναν τουρισμό χωρίς αποκλεισμούς. Ένα πρόγραμμα τουρισμού που δεν θα αποκλείει και δεν θα περιθωριοποιεί κανέναν. Και είναι σημαντικό να ασχοληθούμε με τα θέματα αυτά. Οπότε έχασα ένα μεγάλο τμήμα τη συζήτηση και τον ερωτήσω και σου επαναλάβω κάποια θέματα. Ε, χαίρομαι πάντως που οι μεταφορές στη Φιλανδία είναι σε γυναικεία χέρια. Αυτό είναι πολύ θετικό. Επίσης, ε, κύριε Υπουργέ, μου άρεσε που είπατε ότι θα πρέπει σε αυτήν την νέα εποχή να αναλάβουμε κινδύνους, να φέρουμε τον πολίτη στο επίκεντρο της πολιτικής τουρισμού, του τουρισμού και των μεταφορών. Και επίση επισημάνεται την ανάγκη για συγκεκριμένα αυτά αποτελέσματα προκειμένου να έχουμε ευζοία, ευημερία και μάλιστα βιωσιμότητα αυτής της κατάστασης. Μπράβο σας. Έχω μια ερώτηση για το πακέτο κινητικότητα που φαντάζομαι το αναλύσατε διεξοδικά. Κατάλαβα ότι θέλετε να προχωρήσει το θέμα και ήδη είχαμε τη σχετική θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρόλο που ε, δεν έχουμε καταλήξει ακόμη σε εντολή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις συνδυασμένες μεταφορές, εκεί έχουμε μία κρεμότητα. Επίσης, ε, στα πλαίσια του πακέτου κινητικότητας, ε, τα νοικιασμένα αυτοκίνητα. Ή η ηλεκτρονικη μεταφορά των, των εγγράφων που χρειάζονται για τις επαρωματικές μεταφορές. Σημαντικό θέμα. Και κάτι που δεν αναφέρθηκε μέχρι στιγμής, τα ωράρια. Το Συμβούλιο δεν έχει καταλήξει σε θέση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όμως ψήφισε να καταργηθεί η αλλαγή της ώρας δύο φορές το χρόνο. Εσείς τι γνώμη έχετε για αυτά τα ωράρια, τις, τις δύο αλλαγές της ώρας που γίνονται. Επίση, μιλάμε για τι κλιματικέ αλλαγέ, για του στόχου τη βιομηχανία. Όταν μιλάμε όμω για πολυτροπικότητα, συνδυασμένη χρήση των τρόπων μεταφοράς, ερωτώ, θέλετε να εμπλέξετε τα κράτη-μέλη ώστε επιτέλους να καταλήξουμε σε κάποια σχέδια προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί τα ζητήματα αυτά έχουν κολλήσει λόγω της απροθυμίας των κρατών μελών και αν δεν προχωρήσουμε στα ζητήματα αυτά δεν πρόκειται να υλοποιήσουμε τους στόχους που έχετε. Σας ευχαριστώ. Σας προειδοποιώ ότι το απόγευμα όταν θα σας πω 1,5 λεπτό θα είναι 1,5 και όχι 1,50. και 50. Κυρίες Υπουργέ, βλέπ, υπου, Υπουργοί, συγγνώμη, βλέπετε πόσες ερωτήσεις τέθηκαν για το πακέτο κινητικότητας. Δεν θα κάνω την ιστορική αναδρομή αυτού του πακέτου, το γνωρίζουμε στην Επιτροπή μας, αλλά ο στόχος του είναι σαφής και ξεκάθαρος. Το πακέτο κινητικότητας θα πρέπει να καταλήξει στο να μην έχουμε ε, φορτηγατζίδες εργαζόμενους δεύτερης κατηγορίας. Θέλουμε και για τους ε, οδηγούς των φορτηγών αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά τους. Το ζητούμενο είναι η διασφάλιση της αξιοπρέπειάς τους. Δεν μπορούμε το 2019 να εργαζόμαστε σαν να βρισκόμαστε στις αρχές του αιώνα. Και το πακέτο κινητικότητας έχει δύο σκέλη. Ένα κοινωνικό σκέλος που θα πρέπει να γίνει σεβαστό, αλλά και ένα περιβαλλοντικό σκέλος. Γιατί το θέμα της Ευρωβινιέτας επίσης θα πρέπει να διευθετηθεί. Ένα σημαντικό άλλο θέμα είναι να μεριμνήσουμε ώστε στο μέλλον να καταργηθούν οι καταχρήσεις που διαπράττονται στις οδικές μεταφορές και θέλουμε να σεβαστούμε και τα δικαιώματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά κυρίως θέλουμε να επανενεργοποιήσουμε το θέμα για ίση εργασία, ίσος μισθός, ίση αμοιβή. Και τρίτο ζήτημα για το πακέτο κινητικότητα. Γνωρίζετε κυρίω οι παλιότεροι, οι πιο πεπειραμένοι ευρωβουλευτέ, ότι οι διαπραγματεύσει ήταν χρονοβόρε, διήρκεσαν περίπου δύο χρόνια. Και Σα προειδοποιώ, δεν θέλω να περάσουμε άλλα δύο χρόνια σε διαπραγματεύσεις για το πακέτο κινητικότητα. Φαίνεται ότι και η Φιλανδική Προεδρία είναι πρόθυμη και θέλει να καθοδηγήσει τις διαπραγματεύσεις για να καταλήξουμε σε αίσιο Άλλο σημαντικό θέμα, το κλιματικό. Θα ε, ευχόμουν η Φιλανδική Προεδρία να μας δώσει ένα προσανατολισμό ε, και φιλοδοξίες και στόχους προσιλοποίηση και να ξεκινήσουμε αμέσως στο ειδο... το φύλλο πορείας, τον οδικό χάρτη. Γιατί βρισκόμαστε ήδη στο παραπέντε. Έχουμε 10 χρόνια το πολύ για να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση. Ο χρόνος μας πιέζει, ο χρόνος είναι μετρημένος. Δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου για να αντιμετωπίσουμε τις κλιματικές αλλαγές. Και ε, τα, η προκλήσει είναι τεράστια. Επίση, μεταφορέ. Έχουμε κάποιε περιθωριοποιημένε ζώνε. Έχουμε ε, πρόταση για επαναφορά των νυχτερινών και, ε, τρένων και των ε, δρομολογίων των νυχτερινών με κάποιε πιλωτικέ δράσει που ε, κανένα δεν τι αναφέρει. Επίση, το θέμα τη ουδετερότητα για τι εκπομπές άνθρακα. Πώ θα το επιτύχουμε, Πού είναι ο δικό χάρτη. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Επίση, ναυτιλία να μην ξεχνούμε και τις ναυτιλιακές μεταφορές, τα κρουαζιερόπλια, ο τουρισμός της κρουαζιέρας που αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς. Δεν έχουμε πια κρουαζιερόπλια, έχουμε ολόκληρες πλωτές πολιτείες που δεν σέβονται ούτε τον τοπικό πληθυσμό στις τουριστικές πόλεις όπως είπε η κυρία Ροντρίγκες, δεν σέβονται ούτε ε, την ανάγκη να, προστατευτεί το περιβάλλον και έχουμε πραγματικά ε, τεράστιες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Είπαμε και για την αεροπορία που θα πρέπει επίσης να σέβεται το περιβάλλον. Θα πρέπει λοιπόν να ακούσουμε, να ακούσουμε τις προσδοκίες των πολιτών. Περιβαλλοντικό σκέλος, τι θα γίνει εκεί. Κοινωνικό σκέλος, τι θα γίνει εκεί. Και πώς μπορούν τα τεχνολογικά εργαλεία μας, η ψηφιοποίηση και οι νέες τεχνολογίες να μας βοηθήσουν. Έχετε δύο λεπτά καθεμία παρακαλώ για τις απαντήσεις. Κοίταξια Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολύ καλές ερωτήσεις σας. και για τα σχόλιά σας, τα οποία οπωσδήποτε θα λάβουμε υπόψη στην Προεδρία μας σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαστε εδώ μαζί σας ε, σήμερα και οπωσδήποτε στη διάθεσή σας για να ξαναέρθω στο Κοινοβούλιο να συζητήσουμε αυτά τα σημαντικά ζητήματα. Ο κύριος Ολιβιέ νομίζω επίσης ανέφερε το ότι η προσέγγιση της Φιλανδίας είναι αρκετά ρεαλιστική, τεχνική θα λέγαμε, και η προσέγγιση αυτή από τη σκοπιά του μηχανικού νομίζω φάνηκε και στις ε, παρεμβάσεις μας, αλλά τα παίρνουμε πολύ σοβαρά αυτά τα ζητήματα και θέλουμε να προχωρήσουν. Υπήρχαν πολλές ερωτήσεις για το πακέτο κινητικότητας και βεβαίως θεωρούμε ότι σε μεγάλο βαθμό έχει πάει στους τριμερείς διαλόγους θα ξεκινήσουν κατά τη διάρκεια της ε, προεδρίας μας αλλά πρέπει ακόμα να περιμένουμε ώστε το Κοινοβούλιο να δώσει την διαπραγματευτική του εντολή. Αντιλαμβανόμαστε ότι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο έχουν διαφορετικές απόψεις, οπότε πρέπει να καταλήξουμε σε κάποιους συμβιβασμούς και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να γίνει αυτό. Και αντιλαμβανόμαστε ότι και τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικές απόψεις. Τώρα η κύριοι Ντέλη, Λούντ, Γκριν Λουκασένσα, Λιμπεράτσκι, Νοβακόφ, ήταν Γκραπίνη ρώτησαν επίσης για το θέμα του κοινωνικού πυλώνα. Ο πυλώνας αυτός ε, περιέχει πολλές διαφορετικές απόψεις. Γνωρίζω πως υπάρχουν ευαισθησίες. Ε, όπως είπα εδώ πέρα θα ακούσουμε όλες τις απόψεις ε, όταν ξεκινήσαμε ε, όταν ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις θα δούμε τα πράγματα επακριβώς. Έγινε μια ερώτηση από τον κύριο Μπέρεντ για το διευρωπαϊκό δίκτυο και τα έξυπνα διευρωπαϊκά δίκτυα. Ο στόχος μας εκεί είναι να έχουμε μια γενική προσέγγιση του Συμβουλίου και όπως είπα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσει με το Κοινοβούλιο αν ο χρόνος επιτρέπει. Οι βουλευτέ ε, Λεσαντέ και Λουκασιεύσκα ρώτησαν για τον ε, τομέα της ε, ναυτιλίας και τα κρός Χρειάζεται γρήγορη δράση για να μειώσουμε τις εκπομπέ για να επιτευχθούν οι στόχοι του IMO, του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Και βεβαίως υπάρχουν οι διαφορετικέ απόψει η τεχνολογία και οι αυτοματισμοί προσφέρουν πολλές δυνατότητες για να μειώσουμε τις εκπομπές ε, της ε, ναυτιλίας και πρέπει να συμφωνήσουμε παγκοσμίω για να είναι παγκόσμια σημείο των εκπομπών. Κυρία Τεπερνέ και άλλοι ρώτησαν για τα δικαιώματα των επιβατών σιδηροδρόμων Γνωρίζω πως ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη συμφωνήσει. Ε, είναι κρίσιμο το θέμα, όπως είπα, στόχος Φιλανδίας είναι να υπάρξει μια γενική προσέγγιση του Συμβουλίου τον Σεπτέμβριο, να βρεθεί μια ισορροπημένη λύση όταν ε, μιλάμε για τις υποχρεώσεις των σιδηροδρομικών εταιριών. Μετά, ο κύριος Ντάγγελσον ρώτησε για τις συνδυασμένες μεταφορές και ε, την παρακολούθηση της πρότασης που σχετίζεται με τον ε, πύλωνα της κοινωνικής αγοράς ε, και το πακέτο κινητικότητας. Το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από το πώς θα προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις. Μετά η κυρία Κουταχάρα ρώτησε για την ε, ναυτιλιακή πολιτική και είναι και σχέσεις με τον ΙΜΟ και τα νησιά επίσης. Ε, ο τομέας αυτός είναι πολύ σημαντικός για τη Φιλανδία και βεβαίω ε, θα πρέπει να είναι και σημαντικό τμήμα της πολιτικής των μεταφορών. Δεν υπάρχουν όμως νομοθετικές προτάσεις. Θέλουμε να εστιάσουμε στην συζήτηση για το μέλλον αυτού του τομέα και για τις εξελίξεις στον αυτοματισμό. Η κυρία Βίρκουνεν ρώτησε για το μέσο ενδιόντα στην Ευρώπη και το ΠΔΠ. Όπως είπα, σκοπεύουμε να προωθήσουμε αυτά τα ζητήματα μέχρι το τέλος του έτου, ε, και η οριστικοποίηση τους ε, σχετίζεται με το κατά πόσο θα υπάρξει μια συμφωνία για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και όπως αντιλαμβάνεστε δεν μπορώ να τοποθετηθώ αυτή τη στιγμή για τέτοια ζητήματα και το μέσο ιδιώτα στην Ευρώπη είναι ένα τμήμα αυτή τη υπόθεση. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι το μέσο ιδιώτα στην Ευρώπη και τα διευρωπαϊκά δίκτυα είναι σημαντικά για την εσωτερική αγορά, την περιφερειακή συνοχή. Η κυρία Ροντρίγκε τώρα ρώτησε για τα δικαιώματα επιβατών, αεροπορικών επιβατών. Γνωρίζουμε εδώ πως αυτό είναι σημαντικό θέμα εδώ και καιρό για το Κοινοβούλιο η Φιλανδία θα το επαναφέρει στο επίπεδο των εμπειρογνωμόνων για να συζητηθεί. Σκοπεύουμε να συζητήσουμε την τρέχουσα κατάσταση και το προ ποια κατεύθυνση πρέπει να πάει ο κύριος Ένσλι, όπως και πολλοί άλλοι, αναφέρθηκε στο κλίμα. Όπως είπα, Συμβούλιο Μεταφορών θα γίνει στις 20 Σεπτεμβρίου και θα εστιαστεί αποκλειστικά στο κλίμα, γιατί είναι σαφές ότι οι προκλήσεις αυτές είναι μεγάλες για τον τομέα των μεταφορών, αλλά αποτελούν ταυτόχρονα και μια ευκαιρία. Και είναι βεβαίω σημαντικό να μπορεί να συζητήσει αυτά τα ζητήματα το Συμβούλιο. Ο κ. Φλέγκο ρώτησε για την συνεργασία με την Κροατία, μια χώρα στην ε, τριπλή προεδρία. Έχουμε επαφές ε, ειδικά με την ε, επόμενη Προεδρία της ε, Κροατίας και ακριβώς θα υπάρξει μια συνέχεια στη δουλειά μας. Κυρία μας, ρώτησε για τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Ναι, οι βιώσιμες διασυνδέσεις είναι πολύ σημαντικές, ειδικά για τις μικρές αποστάσεις. Το τρένο είναι μια βιώσιμη δυνατότητα. Δυστυχώς δεν έχουμε πολύ γρήγορο δίκτυο, είναι κατακαιρματισμένο, αλλά για το περιβάλλον είναι σημαντικό να προωθήσουμε ακριβώ τις σιδηροδρομικές διασυνδέσεις. Η κυρία επίσης. Πολλά κρατημέλη δεν έχουν ακόμα υποβάλει τις προτάσεις τους. Κάποια προτείνουν η Κομισιόν να κάνει πιο ακριβείς αναφορές ε, οπωσδήποτε είμαστε σε επαφή με την Κομισιόν και προσπαθούμε να σημειώσουμε πρόοδο. Σας ευχαριστώ τώρα ε, η συνάδελφος για τις ερωτήσεις που αφορούν το δικό της χαρτοφυλάκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις σας. θα απαντήσω στις ερωτήσεις που αφορούν τον τουρισμό. Κύριε Αλέσσοντ, ε, μίλησε για τις κρουαζιέρες και τις περιβαλλοντικές πτυχές. Κοιτάξτε, το 2014 η Κομισιόν έκανε μια ανακοίνωση που αφορούσε ακριβώς ε, την αύξηση της ε, κρουαζιέρας και βεβαίως παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά το πώς εξελίσσονται εκεί τα πράγματα. Πιθανότατα η επόμενη Προεδρία θα δει το θέμα πιο στενά. Και βεβαίως ε, οι κρουαζιέρες ε, σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος ε, και την βιομηχανική πολιτική και την ατζέντα για τη βιώσιμη ανάπτυξη που επίσης αναφέρεται στο πρόγραμμά μας ως προτεραιότητα. Και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η Ευρώπη ε, φτιάχνει στην Ευρώπη να φυγούνται πολλά κροσγερόπλια, πράσινα κροσγερόπλια. Ε, παίζουμε ηγετικό ρόλο εκεί σε αυτόν τον τομέα. Κύριε Στεμπαρνέ και με έτσι ρώτησαν για την οδηγία περί προσβασιμότητας ε, που έχει μεγάλη σημασία και από τη σκοπιά του τουρισμού Στην Προεδρία μας λοιπόν θέλουμε να βελτιώσουμε την προσβασιμότητα διαφόρων σημείων εθελοντικά και να δοθούν οδηγίες στις εταιρείε για να λαμβάνουν υπόψη την προσβασιμότητα. Ανέφερα πριν την ψηφιοποίηση και αυτό έχει σημασία για την βελτίωση της ε, προσβασιμότητας και οπωσδήποτε μπορούμε να αντισταθμίσουμε εν ε, την έλλειψη προσβασιμότητας με την ψηφιοποίηση. Μετά η κυρία Ροντρίγκε Πινιέρο μας ρώτησε για την οικονομία των πλατφορμών, το Airbnb και τα σχετικά Γι' αυτό ακριβώ πρέπει να δούμε τον τομέα τουρισμού, ειδικά στον τομέα της ε, τουριστικής ε, στέγης. Θα υπάρξει μια συζήτηση και... Ο κανονισμός εδώ πέρα αφορά τους υπουργούς εργασίας ε, περισσότερο. Μετά ο κύριος Έινσλι κάνει ένα ερώτημα για την μείωση των εκπομπών και το πώς πρέπει να το δούμε από τη σκοπιά του τουρισμού. Θα ήθελα εδώ πέρα να τονίσω και τον ρόλο της ε, ψηφιοποίησης. Εντάξει, ακούγεται κάπως γενικό και αφηρημένο. Πρόθεσή μας ε, εδώ είναι, αν σκεφτείτε παραδείγματος χάρη, την ανακύκλωση, την πιο, πιο υπηρεσίες, Όλα αυτά είναι τμήμα της ψηφιοποίησης. Και βεβαίως αν δείτε και τους ε, ε κανόνες στην ευρύτερη εικόνα ε, βλέπετε ότι όλα αυτά είναι μια προτεραιότητα του προγράμματος μας. Γι' αυτό ακριβώς αναφέρεται εδώ και η ουδετερότητας προς το κλίμα. Ουσιαστικό κομμάτι εδώ της δουλειά μας. Μετά ο κύριος Φλέγκο ρώτησε για την Προεδρία της Κροατίας. Οπωσδήποτε συνεργαζόμαστε με την Κροατία για να προωθήσουμε και τον βιώσιμο τουρισμό. Έχουμε τονίσει και την ψηφιοποίηση και βεβαίω ε, είναι και δική του προτεραιότητα όταν θα ξεκινήσει η προεδρία τους. Ε, θα ήθελα λοιπόν καταλήγοντας να σας ευχαριστήσω για τις ερωτήσεις σας και τα σχόλιά σας. Ο κύριο Ροχή είπε ότι θα αποστείλει μια επιστολή, οπωσδήποτε το περιμένουμε. Και θα ήθελα να πω πόσο σημαντικό είναι να θυμόμαστε την σημασία του τουρισμού συνολικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας γιατί πολλές ε, τουριστικές επιχειρήσεις είναι μικρομεσαίες και θα έλεγα ότι οι ομάδες εργασίας ε, του Συμβουλίου θα συστήσουν και μια ομάδα εργασία υψηλού επίπεδου και θα έχουμε και το φόρουμ τουρισμού τον Οκτώβριο στο Ελσίνκι. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Ευχαριστώ που μας προσκαλέσατε στην συζήτηση αυτή και εύχομαι κάθε επιτυχία και είμαι σίγουρο ότι θα συνεργαστούμε. Κυρίες Υπουργοί, σας ευχαριστώ και σας ε, σα συγχαίρω διότι η Φιλανδική Προεδρία θέτει ε, ως πρώτη προτεραιότητα την ε, κλιματική αλλαγή. Έχει πολύ καλή θερμοκρασία εδώ στην αίθουσα, αλλά έξω έχει πάνω από 40 βαθμούς στις Βρυξέλλες. Εάν δεν επιταχύνουμε, αύριο δεν θα είναι 40, θα είναι πολύ περισσότεροι βαθμοί. Αυτό σημαίνει ότι όλοι έχουμε ευθύνη οι νέοι μας το ζητούν και δεν μπορούμε να τους κλέψουμε το μέλλον τους. Χρειαζόμαστε ένα καθαρό πλανήτη, αλλά και ένα πλανήτη στον οποίο να μπορούμε να αναπνεύσουμε. Και όταν λέω να αναπνεύσουμε, ένας πλανήτης ε, στον οποίο το θέμα των μεταφορών και ο τουρισμός είναι ε, κομβικά σημεία. Ε, πολύ σωστά απαντήσατε λοιπόν στα θέματα αυτά, θα πρέπει να απαντήσετε για να μας εξηγήσετε πράγματα για την ψηφιοποίηση. Διότι Ποιανού τα δεδομένα, ποιο είναι ο ιδιοκτήτη των δεδομένων. Ο κύριο Έρτουκ αναφέρθηκε στα αυτόνομα οχήνωμα προηγουμένω. Αύριο θα μπορούμε να έχουμε λοιπόν ε, ε, προστασία για τα δεδομένα. Είναι πραγματικό στόχο αυτό. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Είπατε πολύ σωστά ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε και με συγκεκριμένα πράγματα. Συγκεκριμένα πράγματα είναι τα θέματα του προπολογισμού. Είναι να δούμε και τι γίνεται στι νησιωτικέ περιοχέ, τι γίνεται στα νησιά και να μπορέσουμε να διασυνδέσουμε και πάλι κάποιε περιοχέ οι οποίε ορισμένε φορέ είναι ε, απομονωμένοι και ξεχασμένα κυρίω. Και αυτό δεν γίνεται. Επίση, θα πρέπει να μειώσουμε τα αέρια του φαινομένου του θερμοκηπίου με δραστικό τρόπο και ταυτόχρονα να φροντίσουμε να μην λέμε μόνο ότι η οικολογία είναι η μόνη λύση, αλλά υπάρχουν λύσεις. Οι λύσεις είναι πάντα win-win, όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε και τα οικονομικά θέματα, αλλά και το θέμα των πολιτικών επιλογών που πρέπει να γίνουν. Κυρίες μου, ήταν τιμή που σας είχαμε εδώ στην Επιτροπή μου και θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας για το επόμενο εξάμεινο. Ε, θα είμαστε στο πλευρό σας και θα φροντίσουμε αυτός ο χάρτης πορείας να ε, ε, συγκεκριμενοποιηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο για να μπορέσουμε στο τέλος της Φιλανδικής Προεδρίας να έχουμε μια πραγματική επιτυχία μεταξύ των Ευρωπαϊκών Προεδρών. Ε, σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι μπορούμε να σας χειροκροτήσουμε διότι... Exercice pas facile, en tout cas je vous dis à très bientôt. Θα πούμε στο Ιπανεδέν. Η πόρτα του γραφείου μου βεβαίω είναι πάντα ανοιχτή, όχι 24 ώρε το 24 ώρα, όμω, γιατί φεύγω και διακοπέ. Θα τα πούμε σύντομα. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν τελείωσαν οι εργασίε μα. Ε, συνεχίζεται η συνεδρία τη Επιτροπή. Για το επόμενο σημείο, το βρήκα το σφυράκι. Monsieur Liri, vous voulez parler dehors. Όσοι θέλουν να συζητήσουν, σας παρακαλώ εκτός αιθούσης. Tous ceux qui veulent parler, je vous invite à sortir maintenant. Et nous continuons les travaux. Συνεχίζουμε τις εργασίες μας. Θα ήθελα να... Παρακαλώ. C'est la dernière fois. Τελευταία φορά που σας προειδοποιώ. Συνεχίζουμε λοιπόν με το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη για τη μελέτη για τις ε, συνδεδεμένες μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι η τιμή για μένα να έχω εδώ στο πλευρό μου τον ε, συντάκτη αυτής της μελέτης, τον κύριο Ενρίκο Παστόρη. Εσείς θα μας παρουσιάσετε τη μελέτη την οποία έχουμε ζητήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και έχετε 12 λεπτά στη διάθεσή σας για να μας παρουσιάσετε το θέμα αυτό και μετά θα ξεκινήσει η συζήτηση με τους βουλευτές. Έχετε το λόγο για 12 λεπτά. Καλημέρα σας και ευχαριστώ που με καλέσατε να σας παρουσιάσω αυτή την ενδιαφέρουσα μελέτη που ολοκληρώθηκε πέρυσι, αλλά με ιδιαίτερη χαρά θα την παρουσιάσω στην νεοσυσταθήσα Επιτροπή Μεταφορών και ελπίζω να σας χρησιμεύσει και στις μελλοντικές σας συζητήσεις. Ποιο είναι το αντικείμενο της μελέτης. Η παρουσίαση θα ακολουθήσει την ε, δομή της μελέτης. Μία εισαγωγή, μετά κάποια θέματα πολιτικής, μία ανάλυση των δεδομένων, μία, μία παρουσίαση της παρούσας κατάστασης, τα βασικά συμπεράσματα της ε, έκθεσης, βασική φραγμή για, την, για τις συνδυασμένες μεταφορές ή την μετατόπιση προς άλλους τρόπους μεταφοράς και κάποιες συστάσεις. ποιοι είναι οι στόχοι της μελέτης. Να σας παράσχουμε σε εσά και όλους ενδιαφέρομενους μια επίκαιρη και εντελεχή ανάλυση της Προέδρου του Δυναμικού και των, του έργου που έγινε και να εντοπίσουμε ε, τις προκλήσεις που ε, περιλαμβάνονται και στον στη Λευκή Βίβλο του 2011 για τις μεταφορές. Εκεί υπογραμμίζονται κάποιες προκλήσεις και σήμερα θα δούμε και τα, τη μέχρι τώρα πρόοδο που έχει συντελεστεί. Θα επικεντρωθούμε λοιπόν σε κάποια στοιχεία και δεδομένα και θα δούμε μέχρι στιγμής ε, τι σε επετεύχθη. Για να κάνω μια σύντομη ανακεφαλαίωση τη Λευκής Βίβλου για την αλλαγή του τρόπου εκτέλεση των μεταφορών. Αυτό το model shift που λέμε, τι συνδυασμένε μεταφορέ, που είναι στοιχείο τη ευρύτερη στρατηγική, που ξεκίνησε με το στόχο να μειωθεί το διοξείδιο του άνθρακα που παράγεται από τις μεταφορές. Και είναι ένα εργαλείο, αυτό το ανεπίσημο έγγραφο, το white paper, ε, που διευκολύνει την υλοποίηση του στόχου της απαλλαγής από τις εκπομπές άνθρακα. Και για να επιτύχουμε αυτή την απαλλαγή των μεταφορών από τον άνθρακα θα πρέπει να επενδύσουμε στη μετατόπιση προς άλλους τρόπους μεταφοράς. Από τις οδικές μεταφορές δηλαδή προς άλλους τρόπους. Ποιοι είναι οι στόχοι που αναλύσαμε. Καταρχήν 30% ε, μετατόπιση των ε, εμπορευματικών οδικών μεταφορών ε, προς άνω των 300 χιλιόμετρων μέχρι σε προ, πιο βιώσιμους τρόπους μεταφοράς και αυτό θα πρέπει να αυξηθεί το ποσοστό μέχρι το 2050 σε άλλο 30% και για τις ε, επιβατικές μεταφορές μέχρι το 2050 θέλουμε οι περισσότερες ε, μέσεις απόστασης επιβατικές μεταφορές να γίνονται από το σιδηροδρόμους και να τριπλασιάσουμε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Τρένων Υψηλής Ταχύτητας. Αυτό μέχρι το 2050. Ε, πολλές πρωτοβουλίες έχουν ληφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυρίως για όλα αυτά και δόθηκαν διάφορα κονδύλια προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση του στόχου. Αν περάσουμε σε μία ανάλυση των στοιχείων και των δεδομένων που έχουμε, διαπιστώνουμε ότι ε, το μερίδιο ε, της επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές ε, μεταξύ των διαφόρων τρόπων μεταφοράς έχει παραμείνει αμετάβλητο μεταξύ του 1996 και το 2016. Και αν κοιτάξουμε μόνο αυτά τα στοιχεία, διαπιστώνουμε ότι τίποτα δεν έχει γίνει αλλά αυτό δεν ισχύει, δεν αληθεύει, γιατί υπάρχουν περισσότερες διαφορές που είναι ορατές σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Αν δούμε λοιπόν τα στοιχεία σε εθνική βάση, βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα είναι διαφορετικά σε ό,τι αφορά το μερίδιο των διαφόρων τρόπων μεταφοράς στις επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές. Επίσης θα πρέπει να δούμε και τα διάφορα ε, τμήματα, γιατί όταν μιλούμε για τις εμπορευματικές μεταφορές, εκεί ο στόχος ήταν οι εμπορευματικέ μεταφορές ε, σε αποστάσεις άνω των 300 χιλιόμετρων για να έχουμε τη μετατόπιση προς άλλους τρόπους μεταφοράς. Αν δούμε όμως ε, τη ζήτηση για τις σιδηροδρομικές μεταφορές, διαπιστώσαμε την τελευταία δεκαετία μια μεγάλη δυναμική συνδυασμένων μεταφορών, διατροπικών μεταφορών. Ενώ δεν ισχύει κάτι τέτοιο στις εμπορευματικές μεταφορές. Οπότε δεν είναι ίδια τα στοιχεία για τις επερευματικές και τις επιβατικές μεταφορές. Θα πρέπει να δούμε τις τάσεις που ισχύουν στο κάθε, στο κάθε είδος μεταφοράς. Επίσης για τις επιβατικές μεταφορές, όταν βλέπουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις, για παράδειγμα τα τρένα υψηλής ταχύτητας, διαπιστώνουμε ότι χάρη στα τρένα υψηλής ταχύτητας έχουμε μετατόπιση ε, των επιβατικών μεταφορών προς άλλους τρόπους, από τις οδικές δηλαδή προς τις ε, σιδηροδρομικές ή από τις αεροπορικές προς τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Και επίσης δεν θα πρέπει να βλέπουμε μόνο τις μέσες αποστάσεις για τις επιβατικές μεταφορές, αλλά και τις ε, ε υπεραστικές ε, διαδρομές και τις αστικές. Εκεί βλέπουμε σημαντική βελτίωση. Και αν δούμε τώρα τις μελλοντικές ε, προβλέψεις ή τις προσωμιώσεις που γίνονται για το μέλλον, δεν βλέπουμε ιδιαίτερες αλλαγές για το μέλλον. Με βάση το σενάριο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2040-2050, δεν φαίνονται ρηξικέλευθες αλλαγές σε ό,τι αφορά τα μερίδια των διαφόρων τρόπων μεταφοράς. Κυριαρχείων οι ειδικέ μεταφορές. Πώς έχει η κατάσταση τώρα. Η πολυτροπική συνδεσιμότητα είναι βασικό στοιχείο σε περίπτωση που θέλουμε συνδυασμένε μεταφορές. Και υπάρχουν μεγάλες διαφορές στην Ευρώπη. Και υπάρχουν περιοχές όπου η ζήτηση είναι πιο συγκεντρωμένη και πιο μεγάλη για τέτοιου είδους ε, συνδυασμένε μεταφορές. Επίσης, και η ολοκλήρωση των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών δεν είναι ίδια ε, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για το σοδικές σιδηροδρομικές μεταφορές αλλά και το δίκτυο τρένων υψηλής ταχύτητας που απαιτεί τεράστιες επενδύσεις. Εκεί υστερούμε σε σχέση με το βαθμό ολοκλήρωση που περιμέναμε και που είναι χαμηλότερος από τον αναμενόμενο. Επιπλέον ένα βασικό στοιχείο κατά την ανάλυση ε, της ε, έλξης που ασκούν ε, οι σιδηροδρομικές μεταφορές, βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα στη διασυνοριακή διαλειτουργικότητα και συνδεσιμότητα. Δυστυχώς δεν υπάρχει τέτοια διασυνοριακή διαλειτουργικότητα παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει και αυτό δημιουργεί φραγμούς. Πάντω έχει αναλυθεί μια σημαντική πρωτοβουλία που θα αποφέρει καρπούς πιο μακροπρόθεσμα για το θέμα αυτό, για τη βελτίωση τη διασυνοριακή διαλειτουργικότητας. Υπάρχουν όμω και άλλοι λόγοι ε, για τη διαφορετική αυτή συμπεριφορά τη αγορά. Υπάρχουν κάποια κανονιστικά θέματα, για παράδειγμα η χρέωση πρόσβαση των διαφόρων τρόπων μεταφορά. και εκεί είναι διαφορετική πολύ εικόνα μεταξύ των κρατών μελών και για τις οδικές και για τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Εκεί εντοπίσαμε διαφορετικά κριτήρια και διαφορετικά επίπεδα για τα αισθήματα χρέωσης της πρόσβασης. Και κάτι που είναι χρήσιμο και για τις επιβατικές και για τις εμπορευματικές μεταφορές είναι ότι θα πρέπει να εστιάσουμε στις αστικές περιοχές. Εκεί οι δραστηριότητες των αστικών κέντρων αυξάνει τη ζήτηση για επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές. Οπότε στα αστικά κέντρα είναι που λαμβάνονται οι περισσότερες πρωτοβουλίες και εκεί θα πρέπει να επικεντρώσουμε τις δράσεις μας λόγω της αύξησης της ζήτησης. Επίσης, μια καλύτερη ολοκλήρωση μεταξύ των διαφόρων τρόπων μεταφοράς μπορεί να υλοποιηθεί ε, χάρη στην ε, βελτίωση των υποδομών σίγουρα και χάρη στη συμπερίληψη και την ανάπτυξη νέων πολυτροπικών ε, τερματικών και προωθώντας την πολυτροπική συνδεσιμότητα στο θέμα της προσφοράς. Αλλά θα πρέπει να βελτιώσουμε, να βελτιώσουμε και την τεχνολογία με κάποιες εφαρμογές για παράδειγμα. Κοιτώντας τώρα τα αποτελέσματα και την αξιολόγηση, αν δούμε τα δεδομένα, οι στόχοι της Λευκής Βίβλου του 2011 ακόμα απέχουν πολύ από την υλοποίηση. Πιθανώς γιατί ε, είναι και πολύ νωρίς ε, για να μετρήσουμε το αποτέλεσμα αυτό δεδομένου του ότι και η διαθεσιμότητα των υποδομών είναι κάτι το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα να γίνει αυτή η μετάβαση στα άλλα μέσα μεταφοράς και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, θα πρέπει να φτάσουμε μέχρι το 2030 ε, για την επίτευξη αυτού του στόχου. Οι δυνατότητες είναι μεγάλες εκεί όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση της ζήτηση, δηλαδή αστικές περιοχές αλλά και συγκεκριμένες αλλαγές μεταφορών, ειδικά αυτά τα οποία θα πρέπει να μεταφερθούν με συνδυασμένες ε, μεταφορές. Ε, πολλές δυνατότητες επίσης υπάρχουν ακόμα στους ε, σιδηροδρόμους υψηλής ταχύτητας για επιβάτες και βεβαίως οι λοιπές τεχνολογικές εξελίξεις επίσης θα μπορούσαν να ωφελήσουν τη μεταφορά αυτή. Λοιπόν, είπατε 12 λεπτά. Ποια είναι τα βασικά εμπόδια. Αυτό είναι σημαντικό η διαλειτουργικότητα, ήδη είπαμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα διαλειτουργικότητας. Η όρια ανταγωνισμού επίσης είναι ε, κάτι το οποίο ακόμα είναι ζητούμενο. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες ε, για την μελέτη και ανάλυση των εξωτερικών κόστων, του εξωτερικού κόστους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά παρατηρούμε ότι το εξωτερικό κόστος δεν έχει ακόμα εσωτερικοποιηθεί πλήρως, όπως θα έπρεπε, σύμφωνα και με τον στόχο της ε, Κομισιόν, και τέλος η διαφορετική φορολογία των μέσων μεταφοράς και ε, μεταξύ κρατών μελών είναι κάτι το οποίο επηρεάζει κάποια ζητήματα αφορούν την έλλειψη υποδομών, ειδικά για τις πολυτροπικές μεταφορές, ε, έλλειψη προδιαγραφών, ανεπαρκής ανάπτυξη δικτύου σιδηροδρόμων υψηλής ε, ταχύτητας και άλλα προβλήματα, ε, η έλλειψη συντονισμού μεταξύ μεταφορών και χωροταξίας, παραδείγματος χάρη όταν προγραμματίζονται υποδομές ε, παράλληλα με την ανάπτυξη των κέντρων των πόλεων θα μπορούσε να υπάρξει μια συνοχή με την ανάπτυξη ε, των πόλεων όπως είπαμε και βλέπουμε κοιτώντας ειδικά την τεχνολογία πως η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων παροχών ε, στους διάφορους κλάδους είναι ένα βασικό σημείο το οποίο θα βελτίωνε την αποτελεσματικότητα και την ανταγωνιστικότητα του κλάδου. Οπότε ε, έχουμε κάνει και κάποιες συστάσεις εδώ μπορώ να έχω ένα λεπτό. Λοιπόν, οι στόχοι της πολιτικής θα πρέπει να είναι σαφείς και μετρήσιμοι, όπως είπαμε. Π.χ. 300 χιλιόμετρα για τις μεταφορές φορτίου πρέπει να είναι κατομετρήσιμο, γιατί αν δεν έχουμε στατιστικά στοιχεία και συγκρίσιμα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μετρήσουμε αν κάτι έχει επιτευχθεί ή όχι και πιθανώς να καθοριστούν στο στόχοι διαφορετικοί ανά κλάδο μεταφορών. Ο σιδηρόδρομος είναι μεγάλος κλάδος όπως είπαμε αλλά πρέπει να διακρίνουμε μεταξύ συμβατικών μεταφορών που πέφτουν γιατί και η ζήτηση για αγαθά που μεταφέρονται με σιδηρόδρομο μειώνεται ενώ οι διατροπικές μεταφορές, συνδυασμένες μεταφορές αυξάνονται ε, συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Άλλες ε, συστάσεις ε, αφορούν αποτελεσματικά μέτρα για να έχουμε ίσους όρους ανταγωνισμού. Αυτό πρέπει να διασφαλιστεί έτσι ώστε και οι εταιρείε να είναι αποτελεσματικές στην παροχή υπηρεσιών, να επανακαθοριστούν οι προτεραιότητες παρεμάσεων στο δίκτυο, να ενισχύσουμε το δίκτυο εκείνο το οποίο έχει τις περισσότερες δυνατότητες για συνδυασμένες μεταφορές, να επενδύσουμε σε τέρμιναλ συνδυασμένων μεταφορών, το είπαμε, και μετά ε, έχουμε κάποια πιο ήπια μέτρα, δηλαδή την ε, διάχυνση των πληροφοριών, ειδικά στον τομέα των πλεύσιμων ποταμιών, κάτι το οποίο είναι ένα στοιχείο που λείπει, ενώ οι συντηροδρομοί δουλεύουν πάρα πολύ σε αυτό το ζήτημα μέσω των διαδρόμων σιδηροδρομικού φορτίου. Το ίδιο ε, επίσης είναι πολύ σημαντικό ως ανταλλαγή πληροφοριών ε, όσον αφορά τις μεταφορές επιβατών. Θα πρέπει δηλαδή οι χρήστες να ξέρουν ποιες είναι οι δυνατότητες ε, και για να αλλάξουν μεταφορικό μέσο και στο αστικό επίπεδο βλέπουμε τα υφόρα σχέδια αστικής κινητικότητας ε, τα οποία προωθούν πολιτικές για αλλαγή μέσω μεταφοράς και τα λοιπά. Με συγχωρείτε που με Α, αυτά. Είναι μια μεγάλη μελέτη και δύσκολο να την αναπτύξω σε 12 λεπτά. Ευχαριστώ. Σας, Σας ευχαριστώ πολύ. Γι' αυτό ακριβώς ε, και θέλουμε να κάνουμε συζήτηση μαζί σας. Σας ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Αυτό το οποίο... Ή μάλλον να το πω αλλιώς. Διάβασα τη μελέτη σας και έχω πολλά ερωτηματικά. Για παράδειγμα, σε καμία στιγμή στη μελέτη δεν αναφέρεστε στο κόστος ε, το εξωτερικό. Πόσο θα στήχιζε πραγματικά να βρίσκεται κάποιος περισσότερο στο δρόμο παρά για παράδειγμα βάζαμε τα οχήματα ε, πάνω σε ένα τρένο την επομένη. Επίσης, δεν υπάρχει κάτι με το ελεγκτικό συνέδριο που λέει ότι προσέξτε στοιχίζει πάρα πολύ ακριβά ε, να πηγαίνει με τεζεβέ. Ε, επομένως δεν βλέπω κάποιο εφεδρικό στοιχείο στην μελέτη σα και αυτή είναι η πραγματική πρόκληση για τι σιδηροδρομικέ μεταφορές. Αυτό θα μας επιτρέψει την επομένη, την επαύριο να κάνουμε ε, συνδυασμένες μεταφορές. Στη μελέτη αυτή λοιπόν ε, η ανανέωση του σιδηροδρομικού ταμείου θα βοηθήσει. Τρίτη ερώτηση, την οποία επιτρέψτε μου να σας θέσω, είναι ότι ναι, υπήρχε στόχος τον οποίο έπρεπε να προβλέψουμε, ο οποίος δεν είναι υποχρεωτικός, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε και αυτό σε υποχρεωτικό επίπεδο, γιατί το κόστος των ε, σιδηροδρομικών ε, ε, μεταφορών δεν είναι στον κατάλληλη κλίμα. Θα πρέπει να δούμε και τα κλιματικά ζητήματα και επειδή δημιουργούνται θέσεις εργασίας και επομένως θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται με τις εμπειροβηματικές μεταφορές και να επιτύχουμε αυτό το ε, περιβόητο 30%. Πόρο απέχουμε ακόμα. Τι γίνεται επίση με τους μηχανισμούς χρηματοδότηση. Θα πρέπει κάπως να εφαρμοστούν όλα αυτά διότι ακούσατε και τη Φιλανδική Προεδρία. Αναφερθήκαμε στα διάφορα μέσα, στην Ευρωβινιέτα για παράδειγμα. Αυτό θα μπορούσε να είναι χρήσιμο εργαλείο για τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Υπάρχουν λοιπόν πολλά πράγματα. Μπορείτε να μας πείτε πιο συγκεκριμένα λοιπόν σε πόσο χρόνο μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αυτές είναι οι πρώτες μου ερωτήσεις ε, ως πρόεδρος. Και τώρα να δώσω το λόγο σε όποιον θέλει το λόγο. Η κυρία Τάλερ, παρακαλώ. Έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση και για τη μελέτη. Εγώ ως νέος μέλος ε, ε, είναι ένα από τα αναγνώσματα που θα διαβάσω αυτό το καλοκαίρι. Εκ μέρους του ΕΛΚ ε, θα ήθελα να θέσω δύο ερωτήσεις. Η ομάδα μας υποστηρίζει την έννοια της ε, κινητικότητας. Ε, θα ήθελα λοιπόν να προωθήσουμε ολοκληρωμένα συστήματα έκδοσης εισιτηρίων και πληροφοριών ε, στο μέλλον για να βοηθήσουμε την κινητικότητα. Το ρυθμιστικό περιβάλλον βεβαίως θα πρέπει να εγκριθεί εγκαίρως. Τι προτάσεις έχετε να κάνετε εσείς. Και δεύτερη ερώτηση. Εμείς πιστεύουμε ότι η ολοκλήρωση και η διασύνδεση και η διαλειτουργικότητα των ε, μέσων μεταφοράς ε, θα πρέπει ε, να βοηθηθεί και από τις νέες τεχνολογίες, διότι αυτό είναι απαραίτητο στοιχείο των αποδοτικών συνδυασμένων μεταφορών. Έχουμε και φιλόδοξους κλιματικούς στόχους, τους οποίους έχουμε θέσει, να έχουμε μεταφορές με λιγότερη χρήση άνθρακα ε, τι ρεαλιστικού και υπεύθυνου στόχου πιστεύετε θα πρέπει να θέσει κάθε μέσο μεταφορά. Στόχοι που να είναι μετρήσιμοι, διαφοροποιημένοι και να επιτρέψουν να έχουμε ε, αποδοτικές συνδυασμένες μεταφορές. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σέρτουγκ. Όχι, δεν θέλει το λόγο. Ωραία. Η κυρία Μπιλμπάου Μπαραντίκα. Εκτός μικροφώνου, κυρία Μπιλμπάου. Ναι, ήθελα να ευχαριστώ ίσο για τη μελέτη και για την παρουσίαση. Δεν είχα χρόνο ακόμα να αναλύσω όλο το έγγραφο, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω κάτι και να δω μέχρι ναι. ποιο σημείο μπορεί να φτάσουν οι προτάσεις σας. Όντως η Λευκή Βίβλος ε, θέτει πάρα πολλούς στόχους, δεν τους έχουμε επιτύχει και Αναφερόμαστε σε πολλαπλούς τρόπους μεταφοράς, ε, συνδυασμένες μεταφορές, ε, ε, να γίνεται η μεταφορά εμπειροφμάτων με άλλα συστήματα. Αλλά η ραχοκοκαλιά, αυτό το οποίο συζητούμε και ελάχιστα αναφέρουμε και κυρίως για την κλιματική αλλαγή, είναι η κατασκευή των, απα... διευρωπαϊκών δικτύων, που είναι προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως πολύ σωστά είπατε, στοιχίζουν πολλά. Δεν είναι όμως μόνο αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι βάσει των όσων λέει το ηλεκτρικό συνέδριο, έχουν δαπανηθεί πολλά χρήματα, αλλά εξακολουθούμε να έχουμε ένα σύστημα που δεν είναι αποτελεσματικό, είναι κατακαιρματισμένο και το πρόβλημα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει δυνατότητα να υποχρεώσει τα κράτη-μέλη να εκτελέσουν ε, τα έργα εντός προθεσμίας. Τι σημαίνει αυτό αν γίνεται εξωτερική ή εσωτερικοποίηση του κόστους. Αυτό το οποίο δεν αναφέρεται σε καμία έκθεση είναι το πόσο κοστίζει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να κατασκευαστούν, ε, να ολοκληρωθούν μάλλον τα ε, έργα προτεραιότητας, τα οποία έχουν εν μέρη ολοκληρωθεί αλλά δεν είναι πλήρη. Και αυτό που διαπιστώνουμε εδώ είναι ότι η πλειοψηφία των κρατών μελών έχει προβλήματα στα διασυνοριακά κομμάτια, όπου υπάρχει μεγαλύτερο η κυκλοφοριακή συμφέρουση, έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό ε, διοξιδίου του άνθρακα και εκεί έχουμε δει ότι οι οδικές μεταφορές έχουν αυξήσει και τις εκπομπές τους τα τελευταία χρόνια. Τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί αυτό το οποίο μου αρέσει εμένα περισσότερο είναι αυτό το σχέδιο που έχετε όλων των διευρωπαϊκών δικτύων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που σημαίνει ότι αυτό ουσιαστικά είναι το ευρωπαϊκό μετρό και θα πρέπει εκεί να δούμε και το θέμα των, της έκδοσης των εισιτήριων. Εγώ να αγοράζω ένα εισιτήριο στο Μπιλμπάο και να πηγαίνω στο Βερολίνο χωρίς κανένα πρόβλημα. Αλλά δεν μπορώ αυτό να το κάνω. Δεν είμαστε αποτελεσματικοί, δεν χρησιμοποιούμε σωστά τους πέους μας, δεν μπορούμε να καινοτομήσουμε, δεν μπορούμε να μειώσουμε τις εκπομπές, γιατί δεν έχουμε φτιάξει το δίκτυο. Και έχουμε και το ελεγκτικό συνέδριο που λέει ότι δεν είναι για το κόστο, αλλά για το πελατειακό κράτο που ισχύει σε όλε τι χώρε όταν κατασκευάζουν αυτά τα ε, έργα. Πώς μπορούμε λοιπόν να προχωρήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να τα κατασκευάσουμε και να οριστικοποιήσουμε όλα αυτά. Ευχαριστώ. Thank you. Um, Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σίγουρα η έκθεση βρήθη λεπτομεριών και Χαίρομαι γι' αυτό, γιατί πραγματικά θα μας χρησιμεύσει πολύ στη συζήτηση. Με εξέπληξε που δεν δώσατε περισσότερη έμφαση στην ε, ενεργό μεταφορά, όπως θα έλεγα εγώ. Δηλαδή, στο, στην εργασία και την χρήση του ποδηλάτου. Γιατί πραγματικά, ναι. Ε, στο, συγγνώμη, στο, <laughs> στο περπάτημα και στο ποδήλατο. Γιατί πραγματικά αυτή είναι πολύ φιλοπεριβαλλοντική τρόπη μεταφορά και βλέποντας στατιστικές μεταφορές ε, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τα γιοταχή στις ε, μεγάλες πόλεις, όχι μόνο λόγω των καυσέριων, αλλά και στη συμβολή τους στην ποιότητα του αέρα στις πόλεις. Οπότε θα μπορούσαμε να συνδέσουμε την ε, ενεργό μεταφορά με την ανθρώπινη υγεία, γιατί με την αύξηση της ε, παχυσαρκίας. Γιατί να μην συνδυάσουμε στις μεταφορές και την ενεργό μετάβαση στην εργασία με το περπάτημα, με το ποδήλατο, γιατί έτσι θα έχουμε ε, αποσυμφόρηση των οδικών αρτηριών, βελτίωση της ανθρώπινης υγείας, καταπολέμηση παχυσαρκίας. Είναι ένας ε, τρόπος συνδυασμένης μεταφοράς που δεν ε, αναφέρεται καθόλου στην έκθεση. Χαίρομαι που αναφέρετε και το θέμα του φύλου στην έκθεσή σας. Τα τελευταία χρόνια έχουμε πολύ περισσότερη εστίαση σε, στη συμμετοχή και των γυναικών και χαίρομαι που η Εκθεση αναφέρει και το θέμα του φύλου. Είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, μιλήσατε για την υπέρβαση του κόστους στις σιδηροδρομικές μεταφορές. Γιατί δεν αναφέρετε κάτι τέτοιο και στις οδικές μεταφορές, κυρίως σε αυτοκινητοδρόμους. Εκεί δεν υπήρχε υπέρβαση του αρχικού προβλεπόμενου κόστους. Εν λοιπόν, ε, χαιρετίζω την έκθεση. Θα ήθελα μεγαλύτερη έμφαση να δοθεί στο περπάτημα, στο χρήση, στη χρήση ποδηλάτου, γιατί αυτές πραγματικά είναι συνδυασμένες μεταφορές, είναι ενεργός τρόπος μετάβασης από ένα σημείο σε άλλο. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Κουντουρά έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τους συντελεστές της μελέτης αυτής, η οποία παρουσιάζει πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία. Κρατάω καταρχήν από τα συμπεράσματα την, ε, ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει ηγεμονία στις οδικές μεταφορές. Ε, θα ήθελα να σταθώ σε κάποια στοιχεία που παραθέτεται στη μελέτη σας αναφορικά με το σημείο εκκίνησης ορισμένων κρατών, όπως για παράδειγμα σε ορισμένα κράτη οι σιδηρόδρομοι έχουν ε, πολύ χαμηλό ποσοστό διείσδυσης στις μεταφορές εμπορευμάτων ή ακόμα και επιβατών, όπως είναι η Ελλάδα, η Ισπανία αλλά και η Πορτογαλία και η Ιταλία. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις, αν εφαρμοστούν πλήρως οι δικές σας προτάσεις, πόσο θα μπορούσε να αλλάξει το μείγμα μεταφορών τόσο σε εμπορεύματα όσο και σε επιβάτες. Και υποψιάζομαι ότι για να πετύχουμε μια πλήρη ανατροπή του μείγματος και να πιάσουμε τους στόχους μείωσης εκπομπών, μέσω της μεγαλύτερης διείσδυσης των σιδηροδρομικών μεταφορών θα χρειαστούν κάποια μεγάλα ποσά για επενδύσεις σε βασικές ε, υποδομές. Έχετε υπολογίσει τις απαραίτητες επενδύσεις σε βασικές υποδομές. Έχετε προβεί σε μια συγκριτική ανάλυση ώστε να αξιολογήσετε αν υπάρχουν βιώσιμες εναλλακτικέ, όπως παραδείγματος χάρη αυτό που αναφέρθηκε για συνδυασμένες μεταφορές ή ακόμα και για μεγαλύτερη διείσδυση ηλεκτροκίνητων ε, αυτοκινήτων ή φορτηγών. Ευχαριστώ πολύ. Merci, σας ευχαριστούμε κυρία Κουντουρά. Η κυρία Γκραπίνη τώρα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και σας ευχαριστώ που περιλάβατε το σημείο αυτό στην ημερήσια διάταξη και ευχαριστώ που ζητήσαμε εκ μέρους Επιτροπής την ε, κατάρτιση αυτής της μελέτης και ευχαριστώ και του συντάκτε τη. Σίγουρα το περπάτημα είναι σημαντικό, η πεζοπορία, το ποδήλατο είναι σημαντικό, αλλά μην ξεχνούμε ότι οι μεταφορές επηρεάζουν την οικονομία και χρειαζόμαστε μια ανταγωνιστική Ευρώπη στο, στο παγκόσμιο προσκήνιο. Και χαίρομαι που δώσατε έμφαση σε κάποιους τρόπους μεταφοράς που επηρεάζουν την οικονομία. Εγώ είχα εμπειρία στον ιδιωτικό κλάδο και γνωρίζω ποιο είναι το οικονομικό κόστος των μεταφορών. Διατέλεσε και υπουργό της χώρας μου και γνωρίζω τις κλίμακες μεγέθους για το κόστος που συζητούμε. Και σίγουρα υπάρχουν διαφορές μεταξύ εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών. Το θέμα είναι πώς θα αξιοποιήσουμε τη μελέτη σας. Και, και στις δικές μας χώρες κάνουμε μελέτες που καταλήγουν σε κάποια ντουλάπια και δεν χρησιμοποιούνται τα, ε, τα συμπεράσματά τους, δεν αξιοποιούνται οι γνώσεις που προσφέρουν. Πώς μπορούμε λοιπόν να εκμεταλλευτούμε αυτή την μελέτη σας, αυτή την έκθεση, να την αξιοποιήσουμε, σε ποιον να την ε, διαβιβάσουμε, ποιος θα είναι αρμόδιος για την υλοποίηση των στόχων αυτής της μελέτης. Καταφέραμε ε, να βρούμε σημαντικούς δείκτες Λέμε για παράδειγμα ε, για την απόσταση των 20 χιλιόμετρων και κάτω από αυτή να έχουμε εκτροπή των ε, μεταφορών από τις οδικές, ε, από το δικό δίκτυο στις σιδηροδρομικές μεταφορές. Αλλά δυστυχώς έχουμε μεγάλο κατακαιρματισμό του σιδηροδρομικού δικτύου. Δεν έχουμε παντού παρόμοιες υποδομές για τρένα υψηλής ταχύτητας. Και η αγορά είναι κατακαιρματισμένη λόγω του, των διαφορών στις υποδομές. Οπότε, κυρία Πρόεδρε, θα πρέπει η Επιτροπή μας να συζητήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τον επόμενο Επίτροπο Μεταφορών, για να αξιοποιήσουμε αυτή τη μελέτη και να βελτιώσουμε όντως και τους δείκτες. Γιατί αυτό είναι ο στόχος μιας μελέτης. Να καταλήξει σε μετρήσιμους δείκτες και να προτείνει κάποια μέτρα που όταν εφαρμοστούν θα βελτιώσουν την κατάσταση. Ευχαριστώ. Yes, I'm here. Εδώ είμαι. Και ευχαριστώ και για την έκθεσή σας, τη μελέτη σας. Πραγματικά θα είναι ένα ενδιαφέρον ανάγνωσμα για το καλοκαίρι. Έχω μια ερώτηση. Είδα τους πίνακες που μας παρουσιάσατε και είδα και τους πίνακες της τελευταίας 20 ετίας για τις εξελίξεις της μεταφορές. Για κάποιο λόγο, οι εσωτερικές πλωτές μεταφορές δεν αξιοποιούνται πλήρως στην Ευρώπη. Αν δούμε το χάρτη, βλέπουμε ότι υπάρχει σύνδεση από τον Εύξηνο Πόντο προς την άλλη πλευρά της Ευρώπης. Οπότε διαρωτώμε, τι μπορούμε να κάνουμε για να αξιοποιήσουμε καλύτερα τις εσωτερικές πλωτές οδούς και να αξιοποιούμε το Δούναβι για τη μεταφορά εμπορευμάτων, για παράδειγμα. Οι πλωτές μεταφορές, οι εσωτερικές πλωτές μεταφορές είναι και οι λιγότερο δαπανηρές. Είναι πολύ πιο φθηνές από τους άλλους τρόπους μεταφοράς. Και έτσι θα αυξήσουμε και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ε, αγοράς διεθνώς. Να τις αξιοποιήσουμε περισσότερο λοιπόν. Ευχαριστώ. Κύριε Μπλερφέ, λυπάμαι που πριν κατακρεούργησα το όνομά σας με την προφορά μου. Σας ζητώ συγγνώμη. Όλοι αξίζουμε μια δεύτερη ευκαιρία και την αξιοποιήσετε και μπράβο σας, κανένα πρόβλημα. Και ευχαριστώ και τους ερευνητές για την παρουσίαση της μελέτης που μας έκαναν. Ε, η έκθεση δείχνει ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμη μπροστά μας, τεράστιες προκλήσεις. Στα συμπεράσματά σας μιλάτε για, τις, για την εκτροπή των μεταφορών από το οδικό στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Και μάλιστα πήραν τρένα δεν έχουμε πολύ, πολλά τρένα υψηλή ταχύτητα μεταξύ Ολλανδία και Βελγίου. Είναι βέβαια μικρέ οι αποστάσει, αλλά χρειάζονται και εκεί. Επίση, για τι εσωτερικέ πλωτέ οδού, τι δυναμικό υπάρχει, μπορείτε να μα αναλύσετε τι ευκαιρίε και τι δυνατότητε που έχουμε με την εσωτερική ναυσιπλοεία. Γιατί έχουμε εξελίξει και ηλεκτρικού κινητήρε, ηλεκτροκίνητου κινητήρε και για πλοία και στη δημοσιονομική διαδικασία υπάρχει ένα πιλωτικό πρόγραμμα για τη βελτίωση της εσωτερικής ναυσιπλοείας μέσω των εσωτερικών πλωτών οδών των ποταμών. Και περιμένω τα σχετικά αποτελέσματα και τις εκθεσή σας για τα δύο αυτά θέματα. Ο κύριος Φερέιρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον καλεσμένο μας για την παρουσίαση της μελέτης. Δεν πρόλαβα ακόμα να τη διαβάσω. Πάντως, ε, φιλομετρώντας τη πολύ γρήγορα, ε, μου δημιουργήθηκαν ε, δύο-τρεις ερωτήσεις. Πρώτα όμως θα κάνω μια σύσταση γενική. Τέτοιου είδους μελέτες είναι χρήσιμες και πολύ συχνά είναι και ενδιαφέρουσες. Μας βοηθούν στο έργο μας, αλλά δεν είναι ώρα να θετήσουμε μια παλιά καλή πρακτική που είχαμε και αποτυχάσαμε στο μεταξύ και που είναι να μεταφράζουμε σε διάφορες γλώσσες αυτές τις μελέτες και να μην τις έχουμε μόνο σε μία, δύο, τρεις γλώσσες. Παλιά το κάναμε και πραγματικά θα συνέβαλε στην ε, ε, αξιοποίηση και της πολυγλωσσίας και θα μας βοηθούσε και μας το κοινοβουλευτικό μας έργο. Ε, μία ερώτηση που ανακύπτει από τα συμπεράσματα είναι ε, η διαπίστωση ότι τα τελευταία χρόνια είχαμε μια συγκέντρωση των επενδύσεων και της χρηματοδότησης κυρίως σε διασυνοριακά σχέδια και προγράμματα. Αυτός ο προσανατολισμός όμως φαίνεται ότι τίθεται ένα αφιβόλο, Αφισβητείται από μερικούς. Και φαίνεται ότι γίνεται μια προσπάθεια απόσπασης της προσοχής προς μια εθνικά περιορισμένη κινητικότητα ή μια τοπική περιφερειακή κινητικότητα. Αυτό το συμπέρασμά σας μου φαίνεται ενδιαφέρον, μεν, αλλά φοβούμε ότι όλος ο προγραμματισμός που συζητούσαμε μέχρι πρόσφατα και όλοι οι κανονισμοί για τα επενδυτικά και διορθωτικά ταμεία που εξετάσαμε και συζητήσαμε στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία, φοβόμαι ότι δεν είναι προσανατολισμένα όλα αυτά προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Αντίθετα, είμαστε υπερβολικά επικεντρωμένοι στη διασυνοριακή κινητικότητα και αμελούμε τα κενά που υπάρχουν στην τοπική, περιφερειακή, εθνική κινητικότητα. Για παράδειγμα, Είχαμε τον κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Πολύ φοβούμαι όμως ότι η συγκεκριμένη και εύστοχη σύστασή σας δεν αντικατοπτρίζεται στον κανονισμό για τα διαρθρωτικά και παιδιτικά ταμεία. Κάτι άλλο που θα ήθελα να ρωτήσω. Αφορά κάποιες ε, πιθανές συστάσεις της Επιτροπής μας προκειμένου να εγκριθούν κάποια πιλωτικά προγράμματα και προπαρασκευαστικές δράσεις στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί στον τομέα αυτό των συνδυασμένων μεταφορών ή τη μετα... Τη μετατόπιση προ άλλου τρόπου μεταφορά, θα ήταν ενδιαφέρον να έχουμε πιλωτικά προγράμματα και προπαρασκευαστικές πράξει. Και έχουμε κάποιε ήδη προτάσει ε, για πιλωτικά προγράμματα που θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από το κοινοτικό προϋπολογισμό. Γιατί είναι πολύ απεσιόδοξο το σενάριο για την υλοποίηση της, πράσινης, της ε, πράσινης βίβλου για τις μεταφορές. Οπότε μήπως θα έπρεπε να αναζητήσουμε νέους τρόπους ε, για να αλλάξουμε αυτό το σενάριο. Γιατί αν μείνουμε στα γνωστά δεν πρόκειται να υλοποιήσουμε το σενάριο. Ε, τι προτάσεις έχετε λοιπόν ε, για πιλωτικά προγράμματα και παρασκευαστικέ δράσεις ε, που θα μπορούσαν να προκύψουν από την έκθεσή σα και να χρηματοδοτηθούν από το κοινοτικό προπολογισμό. Κύριε Φεραίρα, ο τελευταίο ομιλητή στον κατάλογο, οπότε θα στραφώ και πάλι στον κύριο Παστόρη και θα τον παρακαλέσω να απαντήσει στις ερωτήσεις των συναδέλφων. Α, κύριε Νιούτον, συγγνώμη. Σας ξέχασα. Έχετε και το λόγο. Well, okay. I forgive you. Σα συγχωρώ και εγώ δεν πειράζει. Μια γενική ερώτηση. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Αναρωτιέμαι από τι έρευνε σα τι άποψη αποκομίσατε για την κατάσταση στην Ευρώπη σε σύγκριση με άλλε περιοχέ του κόσμου. Πώ συγκρινόμαστε με την Κίνα, τη ΣΥΠΑ κτλ. Ε, είναι μεγάλη ερώτηση, οπότε ένα γενικό σχόλιο θα ήθελα. Σας ευχαριστώ. Κύριε Παστόρη, Έχετε 10 λεπτά για να απαντήσετε. Ε, παρακαλώ να είστε ακριβείς. Και να μας δώσετε και κάποιες ε, νομοθετικές ιδέες. Εκεί ε, χρησιμεύουν αυτές οι μελέτες ε, για να τις χρησιμοποιούμε μετά συγκεκριμένα στην κατάρτιση της νομοθεσίας. Έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ για τις πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Ε, δεν ήταν εύκολο να απαντήσουμε. Ε, λόγω των διαφόρων θεμάτων. Ξεκινώντας από το τελευταίο, να ξεκινήσουμε από το γενικό, το παγκόσμιο πλαίσιο και να περάσουμε μετά στο ειδικό. δεν κάναμε κάποια σύγκριση με τον υπόλοιπο κόσμο στην ανάλυση αυτή αλλά κοιτώντα ε, τουλάχιστον την ανάπτυξη των υποδομών βλέπουμε τώρα ότι στην Ανατολή, στην Κίνα και σε άλλες χώρες ε, έχουμε γρηγορότερη ανάπτυξη των υποδομών και οπωσδήποτε επενδύουν και σε άλλα μέρη του κόσμου για να βελτιώσουν και να αυξήσουν τις υποδομές και την συνδεσιμότητα των περιοχών πράγματος χάρη αν δούμε τη Βόρεια Αμερική ε, στη ΣΥΠΑ εκεί η κατάσταση είναι ε, ήδη ανεπτυγμένη από το παρελθόν ε, και η κατάσταση ε, ίσως δεν είναι τόσο καλή όσον αφορά τις νέες αναπτυσσόμενες χώρες. Ε, τώρα λοιπόν, κοιτώντας ε, και τις λοιπές ε, υποδομές θα έλεγα πως τώρα εντάξει είναι ένα παράδειγμα εκείνα, αλλά η Ευρώπη είναι πιο περιπλοκό θέμα αυτό το οποίο προτείναμε είναι ε, να μην ξανασκεφτούμε όλες τις στρατηγικές ε, ανάπτυξης ε, υποδομών, απλά να υπάρχουν κάποιες προτεραιότητες. Επενδύσαμε και πρέπει να επενδύσουμε και στο προσεχές μέλλον πολλά λεφτά για την ανάπτυξη των υποδομών και την ολοκλήρωση των υποδομών, που είναι επίσης μια ανάγκη, γιατί Υπάρχουν κάποιοι σύνδεσμοι που λείπουν που πρέπει να ολοκληρωθούν ε, κατά την άποψή μου ε, για να υπάρχει συνέχεια στο δίκτυο. Αλλά πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στις παρεμβάσεις όπου είναι επικεντρωμένη η ζήτηση. Δεν είναι λοιπόν ζήτημα του να μην αναπτύξουμε κάτι διασυνοριακά αλλά οι διασυνοριακές συνδέσει είναι ένα είδος επενδύσεων που κανονικά τα κράτη-μέλη δεν προωθούν. Γι' αυτό ακριβώς ε, θεωρούμε πως και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προωθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση. Όταν μιλάμε τώρα για τις σιδηροδρομικές υποδομές, ε, συζητήσαμε και τη δυνατότητα όχι μόνο ανάπτυξη ε, των σιδηροδρόμων υψηλή ταχύτητας αλλά και το νέο κομμάτι συμβατικών σιδηροδρόμων που τις τελευταίες ε, δεκαετίες ε, έχουν κάπως εγκαταληφθεί σε κάποιες χώρες και άρα και το μοντέλο των τρένων Intercity που υπάρχει στη Γερμανία είναι κάτι το θα μπορούσε να επαναληφθεί και σε άλλες χώρες για να εξοικονομηθούν και χρήματα να μην που θα μπορούσαν να δοθούν σε νέες υποδομές υψηλής ταχύτητας. Και τέλος για να απαντήσω στην ερώτηση για τις οδικές μεταφορές, τις υποδομές οδικών μεταφορών, δεν το εξετάσαμε αυτό. Ε, ήταν εκτός ε, του πεδίου μελέτης γιατί Στόχος ε, της Λευκής Βίβλου ήταν ε, ακριβώς ο τριπλασιασμός ε, του δικτύου τρένων υψηλής ταχύτητα. Γι' αυτό ακριβώς εστιάσαμε σε αυτήν την μελέτη και δεν αναλύσαμε την ανάπτυξη των μεταφορών. Λοιπόν, όταν όμως μιλάμε για την μετατόπιση σε άλλα μέσα μεταφοράς. Ε, αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στην μελέτη. Έχουμε τις υποδομές, ε, τις ε, υπηρεσίες, το πόσο δουλεύουν οι εταιρείες και έχουμε και τους πελάτες. Αυτές είναι τρεις πτυχές πρέπει να δούμε και η ρυθμιστική πτυχή είναι εκεί όπου μπορείτε να παρέμβετε και να δείτε βεβαίως και τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Αυτό λοιπόν όπως είπα στην εισαγωγή μου είναι η βασική πρόκληση της αλλαγής ε, μέσων μεταφοράς, δηλαδή η απομάκρυνση από τον άνθρακα. για να πάμε ακριβώ ε, στους σιδηροδρόμους και πιθανώς ε, και στις ε, υδάτινες μεταφορές που είναι οι πιο φιλικές προς το περιβάλλον. Γιατί αν δείτε τα δεδομένα φαίνεται ότι δεν σημαίνει τίποτα. Αλλά αυτό δεν ισχύει γιατί αν δούμε τις συνδυασμένες μεταφορές αυτές αυξάνονται ειδικά στους πλεύσιμους ποταμούς όπου έχει χαθεί μεγάλος όγκος αλλά είναι η μεταφορά βαρέων αγαθών που πλέον δεν χρειάζεται να μεταφερθούν στα ποτάμια. Και επίσης η καινοτομία, η τεχνολογική, όπως ο εξηλεκτρισμός των αυτοκινήτων, ο εξηλεκτρισμός των πλοίων και των σιδηροδρόμων που έχει ήδη γίνει στο μεγαλύτερο κομμάτι του δικτύου αλλά και η προώθηση ήπιων τρόπων στις αστικές περιοχές είναι όλες δράσεις που οδηγούν στην απομάγνηση από τον άνθρακα των μεταφορών ε, της επιμελητίας. Ε, όλες αυτές οι πρωτοβουλίες ε, λοιπόν μπορούν να βοηθήσουν και μπορούμε και θα έπρεπε κατά την άποψή μου να αναπτύξουμε κάτι προς αυτή η κατεύθυνση. Οπότε για τους πλεύσιμους ε, ποταμούς ε, που ρωτήσατε ε, από, από εκεί για την δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν ο Ρήνος αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται πολύ εντάξει Υπάρχουν κάποιες απειλές που σχετίζονται και με την κλιματική αλλαγή γιατί η στάθμη του ποταμού κάποιες χρονιές είναι χαμηλή και αυτό επιβάλλει κάποιους περιορισμούς στην πλευσιμότητα ενώ εξ όσων γνωρίζω στον Δούναβη δεν ε, υπάρχει ναυσιπλογία σε όλο του το μήκος αλλά υπάρχουν διαφορά κομμάτια του Δούναβη που είναι πλεύσιμα οπότε δεν υπάρχει ε, απευθεία σύνδεση από τη Μαύρη Θάλασσα στην Κεντρική Ευρώπη ε, χρειάζονται λοιπόν κάποιες λύσεις ε, πολλαπλών ε, συνδυασμένων μεταφορών. Τέλος, μια άλλη πτυχή που τονίσατε είναι οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες, όχι μόνο υπηρεσίες, και εκτός εισιτηρίων, κινητικότητα ως υπηρεσία. Αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται, υπάρχει μια έρευνα Βεβαίω, θεωρούμε ότι υπάρχουν πολλές ε, δυνατότητες ε, της ε, πληροφορικής να διευκολύνει την χρήση διαφορετικών μέσων μεταφοράς αλλά δεν είναι αυτή η μόνη πτυχή. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε τις λύσεις πρώτα απ' όλα ώστε η πληροφορική να τις διευκολύνει, να διευκολύνει την μετάδοση και των διαφορετικών πληροφοριών που, πληροφοριών που υπάρχουν στην αγορά, όχι μόνο για τους χρήστες και τους επιβάτες, αλλά για τους χρήστες πολλαπλών μεταφορών, παραδείγματος για την μεταφορά φορτίων. Παρακολουθούμε ότι υπάρχει προσφορά και οι σχετικές εταιρείες προσφέρουν καλές υπηρεσίες, αποτελεσματικές, αλλά κάποιες φορές αυτό δεν ε, ταιριάζει με την ε, ζήτηση των επιχειρήσεων που χρειάζεται να στείλουν τα αγαθά τους ή οι μεταφορείς ε, αγνοούν σε κάποιες περιπτώσεις την ύπαρξη εναλλακτικών πιο φιλικών προς το περιβάλλον. Και μια άλλη πτυχή σημαντική για τις ρυθμιστικές αρχές είναι η ίση του ανταγωνισμού. Συζήτησαμε κάποια ζητήματα στην παρουσίαση. Η Ευρωβινιέτα για τα τέλη κυκλοφορίας είναι κάτι το οποίο συζητάμε εδώ και καιρό ως νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορώ να πω ότι ε, δεν εφαρμόζεται ακόμα Οπότε, εάν η αρχή της Ευρωβινιέτας εφαρμοζόταν, πιθανότατα και η ώρα του ανταγωνισμού θα ήταν πιο ίση από τη σήμερα. Οπότε, όπως είπα στην παρουσίασή μου, και τελειώνω. Υπάρχει μια μακροχρόνια μελέτη για την εσωτερικοποίηση του εξωτερικού κόστους ε, που θα πρέπει να μεταφραστεί σε συγκεκριμένες ε, πράξεις. Ελπίζω να απάντησα στις περισσότερες ερωτήσεις σας. Ε, ίσως όχι σε όλες. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Παστόρη. Η μελέτη σας μας δείχνει ότι έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, γιατί αν πραγματικά θέλουμε να αναλάβουμε την ευρωπαϊκή πρόκληση και σε οικονομικό και σε κλιματικό επίπεδο και χωρίς να ξεχνάμε και έναν από τους τομείς ε, τον οποίο έχουμε ε, μεταχειριστεί πολύ άσχημα είναι ο τομέας των εσωτερικών πλωτών μεταφορών. Ε, μην ξεχνάμε λοιπόν τι ποτάμιε οδού Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ε, διότι δεν τα συζητήσαμε όπω πρέπει, αλλά η Ευρώπη με διάφορου τρόπους μεταφορά ε, δημιουργεί πραγματική ε, διασύνδεση ακόμα και στο τελευταίο χιλιόμετρο. Τα όλα θέματα λοιπόν, επιμελητίας λοιπόν, επιμελητία. Πώ οι πόλεις αύριο θα είναι προετοιμασμένε για αυτή τη μεγάλη πρόκληση τη μεταφορά εμπορευμάτων μέχρι το τελευταίο χιλιόμετρο χιλιόμετρο της πόλης. Ε, όχι να υπάρχουν περισσότερα φορτηγά στις πόλεις, ε, ε, αλλά μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ποδήλατα ή οτιδήποτε άλλο. Τα τελευταία χιλιόμετρα όμως είναι αυτά τα οποία δημιουργούν το τελευταίο πρόβλημα της επιμελητίας των εμπορευμάτων. Θα τη μελετάσουμε τη μελέτη σας κύριε Παστόρη και σας εγγυώμαι ότι θα φροντίσουμε αύριο ε, να δούμε τους στόχους, γιατί αν δεν υπάρχουν στόχοι δεν θα έχουμε ούτε ε, ο, ο, στόχους για το εμπόριο, για πραγματικές επενδύσεις, για διασυνδεμένες μεταφορές. Πρέπει λοιπόν να τα δούμε όλα αυτά. Ε, θέλουμε να έχουμε συγκεκριμένους στόχους και να μπορέσουμε να έχουμε και συνεργασία με τις διάφορες χώρες για να μπορέσουμε να έχουμε και κατάλληλη νομοθεσία. Ευχαριστούμε λοιπόν για την παρουσία σας εδώ και βεβαίως θα σας ε, προσκαλέσουμε και στην Επιτροπή για τις μελλοντικέ ε, ε, εκθέσεις σας μελέτες. Αν έχετε κάποια άλλη ερώτηση για τη μελέτη, μην διστάσετε. Θα τις διαβιβάσουμε στον κύριο Παστόρη για να μπορέσουμε να έχουμε και πιο συγκεκριμένε ερωτήσεις. Δεν συζητήσαμε και τη μέθοδο, διότι η μέθοδος για τις μελέτες είναι πολύ ενδιαφέρουσες ε, γιατί μπορούμε να έχουμε και δυνατότητα σύγκριση, έχουμε μια εικόνα για το τι συμβαίνει στη Γαλλία, τι συμβαίνει στη Σουηδία κλπ. Ο δικό μα ο στόχο είναι να ξέρουμε ε, πού πάνε καλά τα πράγματα, ποιε είναι καλέ πρακτικέ, τι δεν λειτουργεί, για να ξέρουμε ακριβώ ε, τι θα πρέπει να ρυθμίσουμε με συγκεκριμένε λύσει. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ. Ε, θα τα πούμε σύντομα. Συνάδελφοι, καταφέραμε να τελειώσουμε λίγο πιο σύντομα από ό,τι συνήθω. Να σα ευχηθώ καλή όρεξη και θα συνεχίσουμε τι εργασίε μα στι 3. Έχουμε ε, πολύ σημαντική συνεδρίαση. Έχουμε την Επίτροπο Μπούλτς, η οποία θα έρθει σήμερα το απόγευμα για να μας πει... Ε, το επόμενο διάστημα, το οποίο είναι πολύ σύντομο για τη θητεία τη, ε, ποια είναι τα επόμενα σχέδια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Πέρασε στην εθνική.